Θα χρειαστεί να καθυστερήσουμε δυστυχώς ε, μερικά λεπτά ακόμη γιατί πρέπει να εκτυπώσουμε τους καταλόγους των ψηφοφοριών. Πέντε λεπτά καθυστέρηση. Γιατί μία από τις πολιτικές μας ομάδες δεν έχει έτοιμους ακόμα τους καταλόγους ψηφοφοριών. Στο συγγνώμη για την καθυστέρηση. Θα αρχίσουμε το τώρα δυνατό.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 Αρχίσουμε λοιπόν με την έκθεση Τσίμερ ε, για το πρόσωπο της γυναικείας στόχιας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε όλη την ηλεκτρονική σας κάρτα για να δω κι εγώ αν την έχω. Θα είναι πολύ χρήσιμη. Right. Um, amendment... Τροπολογία 5 δεν είναι παραδεκτή. 6 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7 δεν είναι παραδεκτή. Τροπολογία 8 με προφορική τροπολογία που αλλάζει το, τις γυναίκες ε, σε ε, διαμένοντες. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική A, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 10, 11, 12, 13 ε, καταπίπτουν, 14 αποσύρεται, 15 μη παραδεκτή, οπότε πηγαίνουμε στη 16, 17 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται προφορική τροπολογία στο 18 που διαγράφει το, ε, οι περισσότερες εκ των οποίων οι γυναίκες υπέρ, κατά, εγκρίνεται 19 υπέρ, κατά, υπέρ και πάλι, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 20, υπέρ, Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 21 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Απέχετε κυρία Σέκης. Πέραση ψηφοφορία. 18 υπέρ, 11 κατά, 10 αποχές, εγκρίνεται συμβαστική β υπέρ. Μισό λεπτό λέει η πρόεδρος. Καταπέπτει συμβιβαστη... συμβιβαστική β γιατί εγκρίθηκε 22, οπότε περνάμε στην 23. Α, όχι, καταπίπτει και αυτή. 24. Όλα καταπίπτουν, όλες οι τροπολογίες μέχρι... Μισό λεπτό να το βρω. Η 30 έχει αποσυρθεί. μία με προφορική τροπολογία που αλλάζει τις εξής λέξεις ε, των γυναικών και ειδικότερα των ε, ε μόνων γονέων. Υπέρ, κατά, Εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Όχι, να το ελέγξουμε ηλεκτρονικώς, λέει η πρόεδρος. Συγγνώμη. Δεν ε, είδα καλά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. Δεκαέξι υπέρ, 23 κατά, δεν υπάρχουν αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική C, υπέρ. Κατά. Αποχές. 34 καταψηφίστηκε. Λοιπόν, και πάλι ψηφίζουμε. Συμβιβαστική C υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Οπότε, τώρα περνάμε στην 38 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 39 με προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 40 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 41 με την προφορική τροπολογία, το βλέπετε στο έγγραφό σας, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 42 υπέρ, κατά, αποχές, Ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία για την 42. The vote closed. Πέρας ψηφοφορίας. 20 ψήφοι υπέρ, 21 ψήφοι κατά. 20-21 καταπίπτει. Συμβιβαστική D υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στη 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 50 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 51 για διαγραφή υπέρ, κατά, αποχές, καταπίπτει, ε, και απορρίπτεται, συγγνώμη. Ε, συμβαστική ή e υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 53. Ως προσθήκη στη συμβιβαστική e, υπέρ. Κατά. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την 53. Πέρα της ψηφοφορίας. 19 υπέρ, 24 κατά, άρα απορρίπτεται. 56 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 59 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές διαδικαστικό Όχι κατά τη διάρκεια τη ψηφοφορία, συγγνώμη. Εκτός αν μιλάμε, αν είναι για τη συγκεκριμένη ψηφοφορία. Αν είναι δηλαδή για την 59. Προφορική τροπολογία που διαγράφει το εξή, ε, ε, όπου οι γυναίκες ε, απασχολούνται περισσότερο. Αν είναι λοιπόν για το συγκεκριμένο αυτό θέμα, θα δεχθώ το διαδικαστικό. Λοιπόν, 59 υπέρ. Κατά. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την 59.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 έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την 66. one too many I'm from the... Υπάρχει ένας παραπάνω από το ΕΛΚ. Κάποιος να μην ψηφίσει από το ΕΛΚ, παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Και ξαναρχίζει η ψηφοφορία για την τροπολογία 66. Πέρας. Sorry, ψηφοφορία τώρα. Νομίζω ότι τώρα είναι σωστά τα νούμερα. 19 υπέρ, 24 κατά, οπότε απορρίπτεται. 67 υπέρ. Κατά. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την τροπολογία 67. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 36 υπέρ, 7 κατά. Ε, δεν φαίνεται τόσο τσιματσί μας φαινόταν και μία αποχή. Εγκρίνεται. 68. Με προφορική τροπολογία, που το βλέπετε στο εγγραφό σας, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 69 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 70 υπέρ, πάλι με προφορική τροπολογία, υπέρ, κατά, Αποχές. Εγκρίνεται. 71. Υπέρ. Κατά. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την τροπολογία 71. Uh, the vote is closed. Πέρας. 24 υπέρ, 20 κατά, καμία αποχή εγκρίνεται. 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 73 έχει αποσυρθεί, 74 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ κατά Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την τροπολογία 75. Close the vote. Πέρας της ψηφοφορίας. 19 υπέρ, 24 κατά και καμία αποχή. Απορρίπτεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 77 μέχρι 80 έχουν αποσυρθεί. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 82 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 83 έχει αποσυρθεί. Πάμε σε ιδεολογικές σκέψεις. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 2 έχει αποσυρθεί. 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ, κατά, Αποχές. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τελική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Θα ήθελα τότε να θέσω τώρα το διαδικαστικό μου. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με τον κατάλογο ψηφοφοριών στη συμβιβαστική τροπολογία B. Η τροπολογία 23 δεν θα έπρεπε να είχε ψηφιστεί πριν από την συμβιβαστική γιατί δεν επιζητά πλήρη διαγραφή, αλλά μερική διαγραφή. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι η συμβιβαστική B θα έπρεπε να είχε ψηφιστεί πριν από την τροπολογία 22. I'm 22 με ενημερώνουν ότι 22 ε, παρεκκλίνει ακόμη περισσότερο από το αρχικό κείμενο. Γι' αυτό ψηφίστηκε πρώτη. Οπότε περνάμε στην τελική ψηφοφορία, έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. has voted. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. 44 ψήφοι υπέρ, 3 ψήφοι κατά. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια την κυρία Τσίμερ. Διαδικαστικό του κυρίου Σέρκους. Σε σχέση με την συμβαστική θέλω να πω ότι ήθελαν να την υπερψηφίσουν οι σοσιαλιστέ. αλλά κάναμε λάθος που απήχαμε στην 22. Θεωρούμε ότι ήταν συμβατή την B. Ε, Θα ήθελα λοιπόν να καταγραφεί στα πρακτικά ότι η θέση των σοσιαλιστών ήταν υπέρ της συμβαστική B, λέει ο μιλητή. Uh, Καταπίπτει όμως η συμβαστική B εφόσον εγκριθεί η 22. Λυπάμαι γι' αυτό. Ίσως ήταν θέμα με τον κατάλογο των τροπολογιών της ψηφοφορίας. Θα πρέπει να το έχετε θέσει εκ των προτέρων πριν καταρτιστεί ο κατάλογος της ψηφοφορίας. Για τους ελεύθερους το ίδιο μας συνέβη. Έγινε λάθος. Δεν θέλαμε να ψηφίσουμε την 22. Θέλαμε να υπερψηφίσουμε την συμβαστική βή. Ας καταγραφεί λοιπόν στα πρακτικά ότι υπήρξε μια μικρή σύγχυση με την ψηφοφορία. Νομίζω ότι όλοι είχατε την ευκαιρία να δείτε τον κατάλογο των ψηφοφοριών προηγουμένω. Απεστάλησε όλε τι πολιτικέ ομάδε. Ε, κατρίτησαν το δικό του κατάλογο ψηφοφοριών. Τώρα, εφόσον εγκρίθηκε η τροπολογία 22 που ψηφίστηκε πρώτη, ε, κατέπεσε η συμβαστική B. Δεν μπορώ να κάνω κάτι για αυτό τώρα. Και τώρα ψηφίζουμε για την έκθεση της κυρία Χάρκιν. Για το ΕΠ και επέκεινα, ε, καταμέτρηση προόδου σε έναν μεταλλασσόμενο κόσμο. Right, just after I get my tea. Uh, compromise C. Και με το τσάι μου συμβαστική C. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Άρχεται η πληροφορία για την συμβαστική ΣΥ. Πέρας. 24 υπέρ, 18 κατά, εγκρίνεται. Οι υπόλοιπες καταπίπτουν μέχρι την 20. Τροπολογία 20 υπέρ. Κατά. Ψηφίζουμε για την 20 ηλεκτρονικός. Πέρας. 19 υπέρ, 25 κατά. Απορρίπτω. 21 Υπέρ. Κατά. Πάλι θα πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 15 υπέρ, 26 κατά. Απορρίπτεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική D. Υπέρ. Κατά. Θα πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικώς. Συμβαστική D. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 25 υπέρ, 20 κατά. Εγκρίνεται. 23 πίπτη Και φτάνουμε στη συμβαστική ΙΕ. E, Υπέρ. Κατά. Και πάλι θα πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικώς. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. «23 υπέρ, 21 κατά». Εγκρίνεται. Φτάνουμε στην 30 υπέρ. Κατά. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 30. Έχουμε έναν παραπάνω από το ΕΛΚ. Αν μπορούμε να σταματήσουμε και να ξαναρχίσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 30. Πέρας. Υπέρ 23, κατά 18, δύο εποχές. Εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικώς. Άρχεται η ψηφοφορία για την 31. Υπέρ. Με συγχωρείτε. πέρας. 24 υπέρ, 21 κατά. Εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 4. Συμβαστική F. Υπέρ. Κατά. Θα πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικώς. Συμβαστική F, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 26 υπέρ, 20 κατά. Εγκρίνεται. Φτάνουμε με αυτά και με αυτά στη 42. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνατε. 43 υπέρ. Κατά. Θα πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικώς. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 31 υπέρ, 15 κατά. Εγκρίνεται. 44 καταπίπτει. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Καταπίπτει. Συμβαστική G. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Φτάνουμε στην 51. Υπέρ. Κατά. Πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικός Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 19 υπέρ, 27 κατά. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική H υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Φτάνουμε στη συμβαστική I, Ι, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 57 ψηφίζεται ως προσθήκη. 57 υπέρ. Κατά. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικώς και για την 57. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. 19 υπέρ, 27 κατά, καταπίπτει. 60 υπέρ, κατά. Δεν είναι σαφές. Να ψηφίσουμε για την 60. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 19 υπέρ 27 κατά. 61 υπέρ. Κατά. Καταπίπτει. 62 υπέρ. Κατά. Καταπίπτει. Νομι... Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικώς. Άρχεται η ψηφοφορία. Για την 62. Πέρας. 24 υπέρ, 22 κατά. Εγκρίνεται. 63 συμβατεί με την 62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 64 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 65 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 66 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται νομίζω. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική A. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Οπότε φτάνουμε στη συμβαστική J. Στην J, υπέρ. Κατά. Θα πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικώς για την συμβαστική J. Πέρας. 25 υπέρ, 21 κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική K. Κάπα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Θα πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικός. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 15 υπέρ, 27 κατά, ε, απορρίπτεται. Συμβαστική B υπέρ, κατά, αποχές, κρίνεται. Και περνάμε στην τελική ψηφοφορία, διονομαστικής ψηφοφορίας, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 26 υπέρ, 5 κατά, 15 αποχές. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην κυρία Χάρκιν. The final vote is... Τελική ψηφοφορία. Του Ζων Λικβεναμίας για την οδηγία ε, για την εφαρμογή περί Η πρώτη τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 προσθήκη υπέρ κατά θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονική επαλήθευση της τροπολογίας παριθμών 15 παρακαλώ. πέρα της ψηφοφορίας. 18 υπέρ, 26 κατά καταπίπτει, απορρίπτεται μάλλον, η 12 τώρα ως ε, προσθήκη υπέρ, κατά, Απορρίπτεται. 20 κρίνεται απαράδεκτη. Η 21η παρακαλώ, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 22 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 20 Με συγχωρείτε λέει ο Πρόεδρος. Δεζαβίου έχουμε τώρα, μόλις την ψηφίσαμε. Συμβαστική δέλτα, όχι την 22, συμβαστική δέλτα, D δηλαδή, υπέρ. Κατά. Ας γίνει ηλεκτρονική υπαλήθευση παρακαλώ και την συμβαστική D. Πέρας. 22 υπέρ, 21 κατά, δύο αποχές. Εγκρίνεται. 25 τώρα παρακαλώ, υπέρ, κατά, είναι στενά τα ωραία και δεν είμαι σίγουρη ότι έχουν όλοι σηκώσει το χέρι τους. Στην 25 παρακαλώ άρχεται η ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας. 20 υπέρ, 25 κατά, απορρίπτεται. 26 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται με τις ίδιες αναλογίες. 27 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται 32 υπέρ κατά αποχές. Ας επαληθεύσουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά την 32. Δεν ήταν πολύ... Δεν είμαι βέβαιη. Μάλλον ήταν σαφές το αποτέλεσμα, αλλά δεν είμαι βέβαιη. Πολύ σαφέ. 33 υπέρ, 12 κατά. Εγκρίνεται λοιπόν, η 31 πίπτη. η υπαριθμόν 35 καταπίπτει, η υπαριθμόν 33 καταπίπτει, καταπίπτει και η προφορική τροπολογία και προχωρούμε στην 36 υπέρ. Κατά. Δεν βλέπω ακριβώς το αποτέλεσμα, επομένως επαληθεύουμε για άλλη μια φορά με την 36 ηλεκτρονική επαληθεύση. Πέρας προφορές. 29 υπέρ, 15 κατά εγκρίνεται. Τώρα στην 37 παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 38 υπέρ 38 υπέρ. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική ε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Στην 46 θα περάσουμε υπέρ. 46 υπέρ κατά δεν είμαι σίγουρη νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά σε επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά την 46 ε, άρχεται η ψηφοφορία πέρας 24 υπέρ 19 κατά εγκρίνεται η 47 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ κατά δεν είναι πολύ σαφές ας γίνει ηλεκτρονική επαλήθευση για την 48 παρακαλώ άρχεται η ψηφοφορία πέρας 22 υπέρ 20 κατά μία αποχή εγκρίνεται Συμβαστική F, σιγματάφ δηλαδή, υπέρ, κατά. Πάλι δεν σας το αποτέλεσμα. Ψηφίζουμε στη συμβαστική F, άρχιτε ψηφοφορία. Πέρας. 20 υπέρ, 25 κατά, απορρίπτεται. Και έτσι ψηφίζουμε τη 49 υπέρ Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Οι λοιπές καταπίπτουν μέχρι την συμβαστική α. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και περνούμε στην 6 που καταπίπτει εάν έχει εγκριθεί η 14 η οποία δεν έχει εγκριθεί και έτσι ψηφίζουμε την υπαριθμό 6 παρακαλώ, υπέρ, κατά. Και πάλι δεν είναι το αποτέλεσμα, ας κάνουμε την ηλεκτρονική απολύθευση για την 6. Πέρες προφορίες. 23 υπέρ, 21 κατά. Εγκρίνεται η 7 υπέρ. Κατά Ας επαληθεύσουμε όμως την 7 παρακαλώ. Πέρας. 25 υπέρ, 20 κατά. Εγκρίνεται η συμβαστική β υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 10. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται, τελική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία για το σύνολο. Πέρας της ψηφοφορίας. 40 υπέρ. Ε, μία ψήφος κατά, τέσσερις αποχές και συγχαρητήρια στον εισηγητή. together? Uh, we have now two letters on the mobilization of the European globalization agenda. Τώρα έχουμε το θέμα της κινητοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Ψηφίζουμε όλοι μαζί υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ και έτσι ολοκληρώνονται οι ψηφοφορίες. No. Uh, uh, Θα κάνουμε ένα διάλειμμα, πέντε λεπτάκια. Μέχρι να έρθει ο εκπρόσωπο τη Επιτροπή για να συζητήσουμε τα πιλωτικά προγράμματα. Σε πέντε λεπτάκια παρακαλώ να είσαστε όλοι πίσω στην έκθεση. You Σα ενημερώνω ότι απλώς περιμένουμε ακόμη τον εκπρόσωπο της Επιτροπής για τα πιλωτικά προγράμματα. Ελπίζουμε να μην αργήσει. Right, if you'd like to take your seats, please. Thank you. Ε, εντάξει, λοιπόν, αν θέλετε να ξανακαθίσουμε για να συνεχίσουμε. Okay, thank you. Uh, let's get back to uh, the order of business. Ας γυρίσουμε στην ημερήσια διάταξη λοιπόν. Έχουμε την ανταλλαγή απόψεων με εκπροσώπους της Επιτροπής για τα πιλωτικά προγράμματα που εμπίπτουν στο πεδίο των της Επιτροπής Απασχόλησης. Δίνω το λόγο αμέσως στον κύριο Γκίμπερα Μωράου από τη Γενική Διεύθυνση για την Απασχόληση και ήδη έχουμε στις οθόνες την παρουσίασή σας. Thank you, uh, Madam Chair. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Gilbert Μογάν είναι το όνομα του εκπροσώπου της Επιτροπής και αν μου επιτρέπετε θα μιλήσω γαλλικά. Με μεγάλη χαρά έρχομαι να σας παρουσιάσω σήμερα τα συμπεράσματα στα οποία μπορεί η Επιτροπή να καταλήξει ως προς την εφαρμογή των πιλωτικών προγραμμάτων. Έχουμε λίγο χρόνο στη θέση μας και γι' αυτό, κύριε Πρόεδρε, θα πρότεινα να προχωρήσουμε σε δύο χρόνους. Σε πρώτη φάση λοιπόν θα κάνω μια γενική παρουσίαση της θέσης εφαρμογή των πολιτικών προγραμμάτων υπογραμμίζοντας τα διδάγματα τα οποία μπορούμε να κλείσουμε και θα διατυπώσω αν μου επιτρέπετε ορισμένες συστάσεις και επίσης θα απαντήσω σε δεύτερη φάση και στις συγκεκριμένες ερωτήσεις που ενδεχομένω έχουν ε, τα μέλη της Επιτροπής σας για επιμέρους πιλωτικά προγράμματα και αν μου επιτρέπετε επίσης θα ήθελα να από τους συναδέλφους που είναι εδώ σήμερα και με συνοδεύουν να αναλάβουν τις απαντήσεις στις επιμέρους ερωτήσεις για τα πιλωτικά προγράμματα. Ξεκινώ με μία υπενθύμηση ότι σήμερα μιλούμε για οκτώ πιλωτικά προγράμματα με τρία βασικά θέματα το ένα είναι η απασχόληση και η κινητικότητα, το δεύτερο είναι οι συνθήκε απασχόλησης και το τρίτο είναι η προστασία των πιο ευάλωτων. Οκτώ λοιπόν πιλωτικά προγράμματα, εκ των οποίων ε, τα επτά εφαρμόζει η Γενική μας Διεύθυνση και το ε, τελευταίο είναι αυτό της υγείας και του καταναλωτή. Το τελευταίο δηλαδή υπάρχει μόνο οκτώ πιλωτικό πρόγραμμα που έχει να κάνει με τις συνθήκες απασχόλησης στον χώρο της ε, υγείας, στον τομέα της υγείας. Το μέγιστο τμήμα αυτών των ε, πιλωτικών προγραμμάτων με προϋπολογισμό 1 δισεκατομμύριο ευρώ, 1 δισεκατομμύριο ευρώ ε, τέθησε λειτουργία το 2010 αν και δύο από αυτά είχαν ήδη ξεκινήσει το 2008. Το ότι τέθησαν λοιπόν σε λειτουργία το 2010 εν γέννη σημαίνει ότι η Επιτροπή ε, ήδη εφαρμόζει αυτά τα σχέδια και τα περισσότερα από αυτά δεν είναι ακόμη διαθέσιμα ως προς τα λεπτομερή τους αποτελέσματα. Θα μπορούσα δηλαδή σήμερα να παρουσιάσω λεπτομερή αποτελέσματα πιλωτικών σχεδίων τα οποία βρίσκονται εν εξέλιξη. Ε, τα εφαρμόζει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το σύστημα που γνωρίζετε, με, ε, ε, με το σύστημα των προτάσεων και των των προσφορών και τους διαγωνισμούς. Έχουμε το υπαριθμόν τρία πρόγραμμα με την κινητικότητα των εργαζομένων, το οποίο εφαρμόζεται με βάση τις κατευθυντήρες γραμμές EURES, ως προς τα μέσα εφαρμογής, τα εφαρμοστικά μέτρα, και το παριθμόν 4 που έχει να κάνει με την επισφαλή εργασία είναι το μόνο το οποίο θα ε, συνεχιστεί και το 2011 με δύο, με δύο νέες ε, πιστώσεις υποχρεώσεων. Τα λοιπά σταματούν ή συνεχίζονται μόνο με βάση πιστώσεις πληρωμών για το 2011. Στην προσοχή διαφάνεια θα ήθελα να αναφερθώ στην εφαρμογή, τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει τα πιλωτικά προγράμματα. Όπως έλεγα έχουμε να κάνουμε με ε, προτάσεις και προσφορές από τον έξω κόσμο όπως λέμε. Έχουμε λάβει πολλές δηλαδή προτάσεις ως εκ τούτου και ως εκ τούτου και το ποσοστό εκτέλεσης είναι υψηλό για το σύνολο αυτών των πιλωτικών προγραμμάτων. Αν έρχεται περίπου στο 90, φτάνει μέχρι και το 100%. Αν θέλετε λεπτομέρειες στραστικές για κάθε ένα από τα πιλωτικά προγράμματα μπορώ να σας προσφέρω. Πάντως εν γέννη το ποσοστό εκτέλεσης είναι από 90 έως 100%. Με μία μόνο εξαίρεση που θα ήθελα να αναφέρω ρητά και θα επανέλθω κατά τη διάρκεια τη παρουσίαση στο υπαριθμό 3 για την κινητικότητα και την ενσωμάτωση των εργαζομένων, το οποίο όπως είπα εφαρμόστηκε μέσω των κατευθυντηρίων γραμμών Eures και όπου αποδείχθηκε ότι οι μονάδες Eures δεν έχουν αντιληφθεί, δεν αντιλήφθησαν όλες την ευκαιρία που τους προσφερόταν στον τομέα αυτόν. Από τους 49 δικαιούχους ε, δηλαδή Eures μόνο 11 κατέθεσαν προτάσεις για τον τομέα αυτόν με ποσοστό εκτέλεσης αξιοσημείωτα χαμηλό. Είναι δηλαδή κάτω από 20% το ποσοστό εκτέλεσης για το πιλωτικό αυτό πρόγραμμα. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ότι πέραν της ε, επιτυχίες που σημειώνουμε ως προς το ενδιαφέρον των ε, εμπλεκομένων και των δικαιούχων, έχουμε μεγάλο ποσοστό εκτέλεσης όπως είπα και ιδιαίτερα θα ήθελα να επισημάνω στα μέλη τη επιτροπή σα το τι σημαίνει ω προ του ανθρωπινού πόρους σε επίπεδο Επιτροπής διαχείριση αυτών των προγραμμάτων. Άπαξ δηλαδή και υιοθετηθούν τα πιλωτικά προγράμματα μέσα από την ε, δημοσιονομική διαδικασία πρέπει να αναπτυχθεί μια σειρά από ε, βήματα από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποφάσει για την χρηματοδότηση, προετοιμασία, διατύπωση των ε, προσκλήσεων για υποβολή προσφορών, ε, παρακολούθηση της, μέχρι την παρακολούθηση της εκτέλεσης. Στην προσοχή διαφάνεια θα ήθελα σε μια δεύτερη φάση μετά την παρουσίαση εν γέννη των πιλωτικών προγραμμάτων να πω δύο λόγια για την προστιθέμενη αξία και την χρήση των πιλωτικών προγραμμάτων από τη δική μας έποψη. Ένα πρώτο συμπέρασμα λοιπόν, στο οποίο καταλήγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τα πολιτικά προγράμματα, είναι πως είναι χρήσιμα διότι συμβάλλουν στην ανάπτυξη πολιτικών σε επίπεδο και, και ευρωπαϊκό και εθνικό. Είτε πρόκειται για τη συλλογή δεδομένων, προετοιμασία δηλαδή νομοθετικών πρωτοβουλειών, πολιτικών πρωτοβουλειών, και εδώ θα ήθελα να υπογραμμίσω ιδιαίτερως το πιλωτικό σχέδιο για τη συνθήκη εργασία των αποσπασμένων εργαζομένων, με βάση το οποίο θα, γίνουν, θα συλλεγούν στοιχεία τα οποία θα ε, συμπεριληφθούν στην πρόταση τη σχετική για το 2011 και επίσης το, το πολιτικό πρόγραμμα για τη διατήρηση του, της απασχόλησης, της θέσης απασχόλησης που οδηγεί σε μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο του, σε μια πρωτοβουλία για το 2011 πάλι. Άλλο ένα μέσο να συμβάλλουν αυτά τα προγράμματα στην πολιτική έχει να κάνει και με την καλύτερη αντίληψη της κατάστασης, κατανόηση της κατάστασης που επικρατεί στα κράτη-μέλη, στους διαφορούς τομείς και ένα από τα πράγματα που γνωρίζουμε ήδη είναι το εξής, ότι είναι γνωστή η κατάσταση στα κράτη-μέλη ίσως, αλλά μπορούμε να έχουμε περισσότερες πληροφορίες χάρη στα πιλωτικά προγράμματα όπως παραδείγματι, η κακομεταχείριση των ηλικιωμένων ή η πρόσκαιρη απασχόληση ή το ζήτημα των αποσπαστέντων εργαζομένων. Μας δίνουν πιο πολλά στοιχεία λοιπόν αυτά τα προγράμματα και επίσης έχουμε και, το, και την δυνατότητα της ε, ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών όπως για τον αυτισμό, όπως για την ε, κακοποίηση των ηλικιωμένων, τη διατήρηση ε, θέσει εργασία. Τα πιλωτικά προγράμματα έχουν βοηθήσει και στη συλλογή στοιχείων αλλά και στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της κοινωνικής προστασίας και της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Στην προσεχή διαφάνεια θα αναφερθούμε στην ορατότητα την επικοινωνιακή πολιτική, δηλαδή τον απο... σχετική με τα αποτέλεσμα των πολιτικών προγραμμάτων. Καλή βέβαια και η εφαρμογή των πολιτικών προγραμμάτων, αλλά είναι απαραίτητο πιστεύω να εξασφαλίσουμε με πέραν τη συγκεκριμένη εφαρμογή και την ε, κοινοποίησή του στη διάδοση, την ορατότητα δηλαδή αυτών των αποτελεσμάτων και σε ορισμένε περιπτώσει δεν συμβαίνει μεν. Πλην όμω έχουμε μία από τι τρει μεθόδου που σα αναφέρω τώρα, δηλαδή την διάδοση των αποτελεσμάτων μέσω σεμιναρίων που οργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την παρουσίαση αποτελεσμάτων στο πλαίσιο ε, διαφόρων φόρουμ που υπάρχουν, πολιτικών δηλαδή χώρων συζήτησης, Επιτροπή Απασχόλησης, Επιτροπή ε, Κοινωνικής Προστασίας, Επιτροπή ε, Εκπαίδευσης και επίσης τα αποτελέσματα αυτών των πολιτικών προγραμμάτων μερικές φορές εντάσσονται μέσα σε δημοσιεύσεις είτε με τη μορφή μιας μπροσούρας, προσπέκτους, είτε μέσα από το, ε, το, τον διαδικτυακό χώρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και ένα άλλο στοιχείο που θα ήθελα να αναφέρω ως προς την προσθεμένη αξία και την χρήση ή χρησιμότητα των πιλωτικών σχεδίων, για να περάσω στην προηγούμενη διαφάνεια, την υπεριθμών 5, Ένα άλλο στοιχείο προσθέμενης αξίας είναι η προαγωγή των εταιρικών σχέσεων ε, με την κοινωνία των πολιτών. Δηλαδή, σε ορισμένε περιπτώσει, τα, πιλωτικά, τα πιλωτικά προγράμματα είτε συμπεριλαμβάνονται, στα πιλωτικά προγράμματα είτε συμπεριλαμβάνονται, ε, είτε εξ, εξ ολοκλήρου αναλαμβάνουν ιδιώτε, ε, δηλαδή η κοινωνία των πολιτών, και σε ορισμένε περιπτώσει για τρία πιλωτικά προγράμματα, διατήρηση χρόνου αναδιάρθρωση και επισφαλή απασχόληση, τα πιλωτικά προγράμματα εντάσσονται απευθεία σε δράσει που αναπτύσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση τη κρίση. Κρίση που, όπω γνωρίζετε, έχει σαν συνέπεια και την ε, ενίσχυση των επισφαλών, του αριθμού των επισφαλών θέσεων και προβλήματα αναδιάρθρωση κτλ. Και αν μου επιτρέπετε, κυρία Πρόεδρε, θα ολοκληρώσω τη σύντομη παρουσίασή μου με κάποιε συστάσει που ταπεινά σα ζητώ να μου επιτρέψετε να παρουσιάσω στην Επιτροπή σας επί τη βάση των εμπειριών που έχει συλλέξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη λειτουργία αυτών των πολιτικών προγραμμάτων. Έχουμε έξι συγκεκριμένα συστάσει. Η πρώτη σύσταση έχει να κάνει με την ενίσχυση της συνοχής και συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα της Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί μερικέ φορέ διαπιστώνουμε ότι οι δραστηριότητε των πιλωτικών σχεδίων θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από άλλα προγράμματα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό βλέπουμε παραδείγματι στο πιλωτικό σχέδιο για την κινητικότητα μέσω του Γιούρες, την κακομεταχείριση των ηλικιωμένων μέσω του Δάφνη ε, ή τα μέτρα για τη διαφύλαξη της θέσης εργασίας που θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης. Δηλαδή θα πρέπει να προσέχουμε να μην υπάρξει αυτή η επικάλυψη και προκειμένου να αποφύγουμε τον κίνδυνο της υποεκτέλεσης της δημοσιονομικής, διότι στην περίπτωση του Γιούρες έχουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα όπου θα μπορούσε να γίνει χρηματοδότηση από το δίκτυο Γιούρες αυτού του πιλωτικού σχεδίου, το οποίο όμως δίκτυο Γιούρες δεν επέδειξε το απαιτούμενο ενδιαφέρον για την ε, ανάληψη και εκτέλεση του σχεδίου. Η δεύτερη σύσταση, συνδεδεμένη στενά και με την πρώτη, είναι το να εξασφαλίσουμε ότι κατά τον προσδιορισμό των θεμάτων για τα πιλωτικά σχέδια θα ζητείται η γνώμη της Επιτροπής για τα θέματα αυτά, ώστε να υπάρχει και η συμπληρωματικότητα και η συνοχή μεταξύ των πιλωτικών δράσεων και των ε, δράσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τρίτο συμπέρασμα, τρίτη σύσταση, η εστίαση και ο εντοπισμός, ο προσδιορισμός προτεραιοτήτων. Διαπιστώνουμε δηλαδή ότι έχουμε πολλά πιλωτικά προγράμματα με χαμηλή χρηματοδότηση. Τελικά η αποτελεσματικότητα και η προσθέμενη αξία δεν είναι αυτή που θα θέλαμε. Και έτσι προτείνουμε αντί να έχουμε πιλωτικά σχέδια πολυάριθμα με μικρή χρηματοδότηση, να έχουμε λιγότερο αριθμό πιλωτικών σχεδίων, αλλά με πιο σημαντική χρηματοδότηση. Και εδώ, ιδιαίτερα για τον προπολογισμό 2011 που βρίσκεται υπό συζήτηση ακόμα, θέλω να επισημάνω ότι ακριβώ αυτή την προσέγγιση ακολουθήσαμε, γιατί μιλούμε για έναν ε, προπολογισμό 4 εκατομμυρίων ευρώ για το First Job Eures, δηλαδή για την πρώτη θέση εργασία, με βάση το Eures και μετά θα έχουμε ένα ή δύο πιλωτικά σχέδια μόνο που θα συνεχίσει η εκτέλεσή του για το 2011. Έτσι λοιπόν για το 2011 θα έχουμε τέσσερα πιλωτικά σχέδια συνολικά, γιατί έχουμε και εκείνο το οποίο σας ανέφερα νωρίτερα για την επισφαλή απασχόληση. Η τέταρτη μου σύσταση θα ήταν να γίνεται συστηματικά η παρουσίαση των αποτελεσμάτων αυτών των πιλωτικών σχεδίων και των πορισμάτων τους ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συγκεκριμένα της Επιτροπής, όπως έλεγα, βρίσκονται σε ε, στάδιο εφαρμογή αυτά τα πιλωτικά σχέδια. Δεν έχουμε ακόμη συγκεκριμένα αποτελέσματα. Πλην όμως όταν είναι έτοιμα τα αποτελέσματα και τα συμπέρασματα, τα πορίσματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βεβαίω είναι σε θέση για να έρθει και να παρουσιάσει αυτά τα συμπεράσματα. Ένα συγκεκριμένο σχέδιο, πιλωτικό σχέδιο που έχει ολοκληρωθεί πλέον και το οποίο έχει να κάνει με την αναδιάρθρωση και την ε, διαχείριση της βιομηχανικής αλλαγής ε, έχει νομίζω ήδη παρουσιαστεί ενώπιον της Επιτροπής σας. και οι δύο τελευταίες συστάσεις μας, με την αδειά σας, έχουν να κάνουν με την αξιολόγηση, διότι θεωρούμε χρήσιμο, με αυτό το χρόνο, να γίνεται η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των πιλωτικών σχεδίων και των, του αντικτύπου που μπορούν να έχουν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, πράγμα το οποίο από ό,τι γνωρίζουμε ακόμα δεν έχει γίνει. Τελευταία σύσταση να εξασφαλιστεί μια καλύτερη διάδοση των αποτελεσμάτων μέσω των δικαιούχων. Ε, αναφέρθηκα σε μια σειρά από ανακοινώσει δράσεις ανακοινώσεων που έχουν προβλεφθεί. Δεν γίνονται πάντα συστηματικά και θέλαμε να ενισχύσουμε την πτυχή αυτή, κυρίως δηλαδή προσκαλώντα τους δικαιούχου αυτών των ε, σχεδίων ή των επιδοτήσεων να προβλέπουν στο ε, πρόγραμμα, στην προσφορά που υποβάλλουν και την επικοινωνιακή δράση. Μόνο σε μια περίπτωση από ό,τι γνωρίζουμε έχει συμβεί αυτό, δηλαδή στην απασχόληση ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα αυτισμού. Αυτή είναι μια καλή πρακτική που θα θέλαμε να συνεχιστεί και να διαδοθεί ώστε να εφαρμοστεί ευρύτερα και στα λοιπά σχέδια. Ολοκλήρωσα την γενική μου παρουσίαση και θα ήθελα να πω ότι αρχικά προσπάθησα να σας παρουσιάσω τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την εφαρμογή αυτών των πιλωτικών σχεδίων. Στη δεύτερη φάση, όπως είχα πει, τι ε, τις συστάσεις μας. Όπως είπα και πάλι, έχουμε λίγα συγκεκριμένα πορίσματα από αυτή την εκτέλεση των πιλωτικών σχεδίων, γιατί ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί. Πλην όμως, αν θέλετε λεπτομέρειε πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο εκτελεί αυτά τα πιλωτικά σχέδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε εγώ είτε οι συνάδελφοι μας στη θέση σας. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε για την προσοχή σας. Uh, Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμη η παρουσίασή σας. Έχω και εγώ κάποιες ερωτήσεις, αλλά πρώτα θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Η κυρία Μωρέν Σαρτιέ Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ζιλμπέρ Μωράν για την παρουσίαση που μόλις μας έκανε. Είναι ενδιαφέρον, αλλά ούτως ή άλλως κάνουμε μία έκθεση εξέλιξης ε, των διαφόρων σταδίων, ε, όπως άλλωστε είπατε κι εσείς. Ορισμένα στοιχεία που με ενδιαφέραν όλος ιδιαίτερος το τονίσατε κι εσείς, ε, είναι το ποσοστό εκτέλεσης. Όταν βλέπουμε ότι είναι 90, της τάξης του 90 ή 100% το ποσοστό αυτό, πραγματικά πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο ανταποκρίνεται απολύτως στην ε, πραγματικότητα ε, επιτόπου. στις αξιολογήσεις ε, που θα κάνετε και δεδομένου ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το ποσοστό εκτέλεσης των προγραμμάτων, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσετε παράλληλα να παρακολουθήσετε τον αντίκτυπο των προγραμμάτων και του ποσοστού εκτέλεσής τους σε άλλα κλασικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, υπήρχαν ε, φαινόμενα ε, μεταφοράς, δηλαδή ε, υπήρχαν ας πούμε περισσότερα πυροτικά προγράμματα αλλά λιγότερες δραστηριότητες ε, στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων που ομοιάζουν με τα προγράμματα που έχουν σημαντικό ποσοστό εκτέλεσης. Είναι πολύ σημαντικός λοιπόν αυτός ο συσχετισμός και είναι ένα ζήτημα για το οποίο εμένα τουλάχιστον θα με ενδιέφερε να γνωρίζω περισσότερα. Δεύτερο σημείο που μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον είναι η αξιολόγηση του πραγματικού αντικτύπου στις εθνικές πολιτικές. Δηλαδή, θα υπάρξει νέα νομοθεσία, θα υπάρξουν ε, εθνικά προγράμματα τα οποία θα συνεχίσουν αυτή την προσπάθεια των ευρωπαϊκών ε, πιλωτικών προγραμμάτων. Θα είναι δηλαδή πραγματικά τα πιλωτικά αυτά προγράμματα πηγή έμπνευσης ε, για περαιτέρω εθνικά προγράμματα. Αυτή τη στιγμή ολοκληρωθούν τα πιλωτικά. Αυτά λοιπόν είναι δύο ζητήματα επί των οποίων πιστεύω ότι πρέπει να εστιαστούμε. Και το τρίτο θέμα που θα ήθελα να θίξω, οι δικαιούχοι Ε, ε, είναι, είναι πραγματική η ε, ορατότητα των προγραμμάτων αυτών ως προγράμματα ευρωπαϊκά. Δηλαδή, εμείς όταν πηγαίνουμε επί τόπου βλέπουμε ότι όταν υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα πολλά πολιτικά, όπως για παράδειγμα η πολιτική για όσους... για τους αυτιστικούς, για παράδειγμα είναι ε, πραγματικά κατανοητά σε τοπικό επίπεδο, μήπως ε, μπορούμε να τα καταστήσουμε ακόμη πιο κατανοητά, ακόμη πιο σαφή για τους ε, συμπολίτες μας. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Σρότερ και μετά ο κύριος Κρίστενσεν. Θα ήθελα να για την περίπτωση που αναφέρατε για το Γιούρες που δεν ε, πήγε καλά. Είναι βέβαια αυτό, αλλά και άλλα σχέδια τα οποία αναπτύσσονται σε συνεννόηση, τη συνεργασία με τους χειρονικούς εταίρους. Αυτό που δεν θέλω εγώ να μάθω, και έχω καταθέσει και τη σχετική ερώτηση ως βουλευτής, οφείλεται αυτό στην Επιτροπή και τον τρόπο με τον οποίο έχουν περιγραφεί αυτή η όροι. Γιατί πιστεύω ότι αυτό έχει συμβεί και είναι κρίμα γιατί πρόκειται για πολύ σημαντικά σχέδια. Σχέδια τα οποία είχαν αποφασιστεί να εκτελεστούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το 2004-883. Είναι λυπηρό το ότι δεν είναι ικανοποιητικά τα αποτελέσματα και εκεί που μιλήσατε εσείς για τη συνοχή και την ε, προσαρμογή στις κατάλληλες γραμμές του προϋπολογισμού, βλέπω ότι έχετε λησμονήσει στη συνοχή ένα πολύ σημαντικό θέμα, αυτό που έχει να κάνει με τα τρόμενα αναπηρίες. Αυτό πώς εξηγείται. Ο κύριος Κρίστενσεν, ευχαριστώ πολύ και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρουσίασή του. Είναι πάρα πολύ, σημαντικό πόσο διαμεσολαβητικό ρόλο παίζουν αυτά τα προγράμματα. Και νομίζω ότι είναι και αρκετά σημαντικός δείκτης ε, του πώς, του πόση πρόοδο σημειώνεται στο πλαίσιο, για παράδειγμα, των κοινωνικών ταμείων. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς ένα πιλωτικό πρόγραμμα μπορεί να επηρεάσει την κατάσταση σε άλλες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι επαρκές να έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Επιτροπή μας όταν έχουν ολοκληρωθεί τα προγράμματα ε, και μόνο. Νομίζω ότι πρέπει να γνωρίζουμε περισσότερα πράγματα και κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων, κατά την εξέλιξή τους. το να λέμε απλώς ότι δεν χρειαζόμαστε περαιτέρω πιστώσεις για κάποια ε, προγράμματα... Είναι ενδιαφέρον, αλλά είναι ενδιαφέρον να ξέρουμε ότι στο πλαίσιο μια συγκεκριμένη χρηματοδότητα είναι ενδιαφέρον να κάνουμε και άλλα πράγματα. Γιατί μια τέτοια αξιολόγηση, αφού έχει ολοκληρωθεί ένα πρόγραμμα, δεν έχει πάρα πολύ νόημα γιατί δεν, έχει πολύ, δεν έχουμε ε, τη δυνατότητα να, συμπεριληφθεί, να συμπεριληφθούν επιπλέον πιστώσει στον προϋπολογισμό. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω να έχουμε και μία αξιολόγηση κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν πλήρες επιστώσεις ε, του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Εκούς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω, όπως και οι συνάδελφοι, για την παρουσίαση των υπεύθυνων της Επιτροπής. Ελπίζω ότι θα λάβουμε και αντίγραφα. Και ήθελα με κάθε ευγένεια βέβαια να πω ότι δεν είμαι πλήρως ικανοποιημένους. Γιατί παρόλο που είχαμε μια παρουσίαση για τις προπαρασκευαστικές δράσεις των πιλωτικών προγραμμάτων του 2010, δεν είχαμε συμπληρωματικές πληροφορίες σήμερα το πρωί. Δηλαδή, υπάρχουν πιλωτικά προγράμματα και προπαρασκευαστικές δράσεις που τρέχουν εδώ και 30 χρόνια. Και για την ώρα έχουμε μόνο μια πολύ επιφανειακή ενημέρωση για το τι ακριβώς συμβαίνει. Είδαμε κάποιες περιπτώσεις που πετυχαίνουν όπως στα μικροοικονομικά όπου πολλές διαφορετικές πολιτικές θεσπίστηκαν ε, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως κατά τη δική μου την αντίληψη της παρουσίασης της Επιτροπής σήμερα το πρωί, τα πιλωτικά προγράμματα είναι βάση για την λήψη αποφάσεων, δεν είναι μάλλον βάση αποφάσεων για και για, το, για την, ε, σχεδιασμό νέων δραστηριοτήτων στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απλώ οδηγούν στη διοργάνωση εσωτερικών συναντήσεων στην Επιτροπή και εσωτερικού συντονισμού. Ε, για του δημοσιονομικού μα λοιπόν πόρου και την παραδοσιακή στήριξη που δίνεται από το Ευρωκοινοβούλιο στα πιλωτικά προγράμματα, είναι σημαντικό να ε, ξεπεράσουμε την διοικητική αδράνεια που φαίνεται να επικρατεί. Θα πρέπει δηλαδή να δούμε κατά πόσον γίνονται, μπορούν να γίνουν τα, πολιτικά προγράμματα πιο εύστοχα ως προς το γενικό σχεδιασμό μας πολιτικής. Πρέπει να είμαστε λοιπόν πολύ προσεκτικοί στην αξιολόγηση του τελικού σκοπού, της τελικής χρήσης των πιλωτικών προγραμμάτων. Οι πραγματικές καινοτόμες δράσεις που προβλέπονται στις πολιτικές των ε, κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι αυτές που θα πρέπει να μας καθοδηγούν. Γι' αυτό με ικανοποιούν ιδιαίτερως οι συστάσεις, οι έξι συστάσεις που ακούσαμε, διότι μπορούν να αξιοποιηθούν έτσι ώστε στην επόμενη συνάντηση που θα έχουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχουμε, ελπίζουμε, ένα καλύτερο πλαίσιο αξιολόγησης. Κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να δούμε σε τι βαθμό τα πιλωτικά προγράμματα μπορούν να χρησιμοποιούνται για να χρησιμοποιηθούν ω βάση σχεδιασμού νέων πολιτικών. Και το Ευρωκοινοβούλιο βεβαίω θα πρέπει να τηρείται ενήμερο. Αλλά θα πρέπει και να μπορούμε να ελέγχουμε τα αποτελέσματα των πιλωτικών προγραμμάτων. Ήθελα να θέσω και ένα ερώτημα προ τον εκπρόσωπο τη Επιτροπή. Δηλαδή, πώ μπορούμε συστηματικά να ενημερωνόμαστε Πώ θα μπορούσε να ενισχυθεί αυτή η σχέση συνεργασία μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου και Επιτροπή, ώστε να βλέπουμε την κάθε μια από τι προπαρασκευαστικέ δράσει και τα πιλωτικά προγράμματα και πώ ακριβώ υλοποιούνται. Ευχαριστώ. Απλώ να ενημερώσω του συναδέλφου ότι υπάρχει έγγραφο στο φακέλου σα, λογικά το έχετε λάβει ήδη, για τα πιλωτικά προγράμματα του 2011 και τι προπαρασκευαστικέ του δράσει. Είναι πολύ χρήσιμο, αλλά θα αποστείλουμε αντίγραφο και με email σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Ήταν πολύ χρήσιμη. Αλλά λαμβάνοντα αφορμή των σχολείων κάποιων από τους συναδέλφους. Για αυτά που είπατε κι εσείς ο ίδιος. Για την πληροφόρηση. Ξέρετε, έχετε εσείς ο ίδιος κάποια προσωπική άποψη για το πώς μπορεί να βελτιωθεί αυτή η διάδοση των πληροφοριών. Μιλήσατε για τους συνομιλητές, τους εταίρους που θα πρέπει να έχουν και ενεργό συμμετοχή στα σχεδιασμό των πιλωτικών προγραμμάτων. Όμω αυτό που είπε η κυρία Μωρά Σαρτιέ, ε, πώ μπορούμε να διαδίδουμε καλύτερα αυτέ τι πληροφορίε στα ίδια τα κατημέλη, πώ μπορούμε να περνάμε το μήνυμα, ώστε τα πολιτικά προγράμματα λόγω χάρη να μην ε, την χάνουν καταχρήσεων. Ε, είπατε ότι υπάρχει εδώ μια επικάλυψη μεταξύ κάποιων προγραμμάτων. Μπορείτε να επεκταθείτε λιγάκι στο τι γίνεται ας πούμε, με την κακομεταχείριση των ηλικιωμένων και τα σχετικά πιλωτικά προγράμματα. Τι είδου συσχετισμό υπάρχει μεταξύ των όσων κάνετε εσείς και στο πρόγραμμα Δάφνη για, το, ε, για να περιοριστεί η κακομεταχείριση των ηλικιωμένων. Τι ακριβώς συμβαίνει σε σχέση με άλλου τομείς. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να καταλάβουμε πώ όλα αυτά συσχετίζονται. Εάν μπορούμε να έχουμε έναν αποτελεσματικότερο τρόπο να δρούμε. Και αποτελεσματικότερο τρόπο να προβάλλουμε αυτές τις πληροφορίες ώστε τα κράτη-μέλη όταν σχεδιάζουν τις πολιτικές τους να μην χρειάζεται τότε να χάνουν χρόνο και να κάνουν την έρευνα εκείνη τη στιγμή. Συχνά μιλώ με ανθρώπους που λένε ότι χρειαζόμαστε περισσότερη έρευνα, περισσότερες μελέτες. Και αναγκάζομαι να του πω ότι μα έχει γίνει αυτή η μελέτη και να του υποδείξω την κατεύθυνση που θα την αναζητήσουν. Εάν λοιπόν κάποιο από εσά έχει επιπλέον στοιχεία για το πώ μπορεί να διαδίδεται αυτή η πληροφορία, αυτέ οι πληροφορίε, θα ήταν ε, άκρο χρήσιμο. Σα δίνω και πάλι το λόγο σε εσά ή στου συναδέλφου σα για να απαντήσετε στα ερωτήματα. Um, thank you, um, madam. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στα ερωτήματα τουλάχιστον τα γενικά, και θα ζητήσω από του συναδέλφου να δώσουν ειδικότερε απαντήσει στα συγκεκριμένα προγράμματα. Λόγω χάρη για το ερώτημα τη κυρία Σέτερα για το Γιούρες, το πιλωτικό πρόγραμμα Γιούρες. Πρώτα απ' όλα, να θυμίσω ότι μιλάμε για προγράμματα σχετικά μικρή κλίμακα. Πιλωτικά προγράμματα περίπου του 1 εκατομμυρίου ευρώ τα οποία πολλές φορές καλύπτουν όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε μιλούμε για μικρά προγράμματα. Και για να είμαι ειλικρινής, ε, είναι ανάλογος και αντίκτυπος. Δηλαδή, ένα πιλωτικό πρόγραμμα ενός εκατομμυρίου σε όλα τα κράτη-μέλη είναι ένα, ένα πολύ μικρό αποτέλεσμα για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό ακριβώ συστήνουμε να έχουμε λιγότερα πιλωτικά προγράμματα αλλά μεγαλύτερου μεγέθους. Έπειτα, για την αξιολόγηση. Επεσήμανα στην παρουσίασή μου και το λέω για τους συναδέλφους σας, τον κύριο Σέρκας και την κυρία Μωράν Σαρτιέ, ότι η σημασία αξιολόγησης των πολιτικών προγραμμάτων εκ των προτέρων και εκ των υστέρων είναι κάτι που δεν γινόταν στο παρελθόν και να σας πω γιατί. Ε, πρέπει να αξιολογούμε τον αντίκτυπο των πιλωτικών προγραμμάτων και θα μπορούσαμε να αξιολογούμε αυτόν τον αντίκτυπο με διάφορους τρόπους, όμως το πώς επηρεάστηκε η πορεία των πολιτικών των κρατών μελών από τα πιλωτικά προγράμματα, πώς αναπτύχθηκε η πολιτική των κρατομέλων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, Πώ υλοποιήθηκαν τα πιλωτικά προγράμματα σε κάποιε περιπτώσει σε σχέση με τι πολιτικέ ή άλλα προγράμματα που έτρεχαν παράλληλα, εάν υπήρξαν επικαλύψεις και αν όχι γιατί, όλα αυτά είναι ένα φάσμα στοιχείων, υπάρχει ένα πεδίο το οποίο πρέπει να μελετήσουμε και να διερευνήσουμε και με μεγάλη μας χαρά θα το κάνουμε σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Επίσης συμφωνώ ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε την ε, συνεργασία, το συντονισμό με άλλα παράλληλα προγράμματα. Κάτι που είπε και η κυρία Μωράν Σαρτιέ και εσείς, Πρόεδρε. Είναι σημαντικό εδώ. Πιστεύω ότι γενικώ τα πολιτικά προγράμματα συμπληρώνουν όσα κάνουμε μέσω άλλων προγραμμάτων. Στο βαθμό του δυνατού εξασφαλίζουμε τη συμπληρωματικότητα μεταξύ πολιτικών προγραμμάτων και των ε, προγραμμάτων που ήδη εφαρμόζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα πιλωτικά λοιπόν προγράμματα πρέπει να εξυπηρετούν το σκοπό τους και δεν θα πρέπει να παρεκκλίνουν τελείως από αυτόν. Όμως, όπως είπα, υπάρχει και περίπτωση γιούρες, όπου κάτι τέτοιο δεν συνέβη δυστυχώς. Επίσης συμφωνώ ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε την προβολή των πιλωτικών προγραμμάτων. Στο βαθμό του δυνατού βεβαίω, αλλά ούτω ή άλλω μην ξεχνάμε ότι είναι μικρή εμβέλεια προγράμματα. Θα ήταν λοιπόν χρήσιμο να ακούσουμε και τον ε, συνάδελφό μου, ε, εξ τον κύριο Λεμπρά, για την ε, τεράστια προσπάθεια διάδοση που έχει γίνει σχετικά με τα πιλωτικά προγράμματα και την αναδιάρθρωσή του. Ένα πολύ καλό παράδειγμα του είδου προβολή και επικοινωνία που πρέπει να διοργανώσουμε. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό για τα αποτελέσματα των πιλωτικών προγραμμάτων και θα σας εξηγήσουν οι συνάδελφοι για το συγκεκριμένο πιλωτικό πρόγραμμα πώς παρουσιάστηκε στην άτυπη ΕΠΣΚΟ στην Ισπανία στους υπουργού. Δηλαδή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κοινωνικών Υποθέσεων. Ένα πολύ καλό παράδειγμα λοιπόν καλών πρακτικών. Θα συμφωνήσω και με του ε, βουλευτέ που είπαν ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε την ε, τακτική ενημέρωση αυτή τη Επιτροπή για την εξέλιξη των πιλωτικών προγραμμάτων και να μην έχουμε μία ε, μεμονωμένη παρουσίαση όπως η σημερινή. Πρέπει να υπάρχει μια συστηματική παρακολούθηση του τι γίνεται. Αυτό πιστεύω ότι θα εξυπηρετήσει καλύτερα το σκοπό ενημέρωση του Κοινοβουλίου σε, σε τακτά χρονικά διαστήματα. Και τέτοια ανταλλαγή απόψεων δεν έχει να κάνει μόνο με τη δική σας την ενημέρωση για τα πιλωτικά προγράμματα, αλλά και για να γίνει συζήτηση μαζί σας για το κατά πόσον πρέπει να συνεχίσουν κάποια πράγματα ή όχι. Ιδανικά μια τέτοια συζήτηση πρέπει να γίνεται όταν εσείς συζητάτε στην Επιτροπή σας τα πιλωτικά προγράμματα. Οπότε θα, θα μπορούσατε να, προκα... να προσκαλείτε τότε την Επιτροπή ώστε να σας πει τα δικά της τα στοιχεία ποια είναι για τα συγκεκριμένα πιλωτικά προγράμματα. Τα μελλοντικά και επευκαιρία τα εξελισσόμενα ως προς την ε, συμπληρωματικότητά τους και την ε, συμβατότητά τους. Έτσι όπως εφαρμόζονται και υλοποιούνται από την Επιτροπή. Μια από τις παρατηρήσεις σας, Πρόεδρε, <clears throat> για τη διάδοση των πληροφοριών. Όπως είπα, Έχουμε καλά παραδείγματα, θα σας τα πούνε τόσο λίγο οι συνάδελφοι, για την επιτυχή διάδοση. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό Δηλαδή θα έπρεπε ενδεχομένω να υπάρχουν προγράμματα, μάλλον στοιχεία επικοινωνία ε, που να συμπεριλαμβάνονται ήδη στα πολιτικά προγράμματα τα ίδια. Να είναι ενσωματωμένα. Ένα σχέδιο επικοινωνία, προβολή, ώστε οι δικαιούχοι να ξέρουν ε, εκ των προτέρων ότι η προβολή των αποτελεσμάτων, η διάδοση των πληροφοριών είναι από τα στοιχεία τη υλοποίηση του πολιτικού προγράμματο. So in a nutshell, um, I Εν ολίγης, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Μπορούμε να βελτιώσουμε τη διάδοση, να έχουμε μεγαλύτερη προβολή των αποτελεσμάτων και υπάρχουν ήδη καλά παραδείγματα τέτοιων προσπαθειών. Απλώς το ποσοστό εκτέλεσης δείχνει ότι υπάρχει ζήτηση για τέτοια προγράμματα και σε πολλές περιπτώσεις έχουμε περισσότερα προγράμματα από ότι επέτρεπουν ενδεχομένως τέτοια τα προγράμματα. Το θέμα είναι ότι με τον περιορισμένο αυτό αριθμό προγραμμάτων ούτω ή άλλω δεν φτάνουν οι πόροι. Και να επανέλθω στην αρχική μου παρατηρήση που νομίζω ότι είναι καθοριστική σημασία. Αν θέλουμε να είναι αποτελεσματικά τα πιλωτικά προγράμματα και να έχουν αντίκτυπο στην πράξη, θα πρέπει και πάλι. Και το τονίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε λιγότερα προγράμματα, με μεγαλύτερο προπολογισμό ωστόσο. Και αν μου επιτρέπετε, Πρόεδρε, να δώσω τώρα το λόγο στο Ζων Φρανσουά για το θέμα της διάδοσης και στον κύριο Κομφέρη για το Γιούρες. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. θα σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα της ε, διάδοσης των πληροφοριών ε, για πιλωτικό πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει από το 2008 σε σχέση με την ε, βοήθεια προς τους εργαζομένους κατά τη διάρκεια της αναδιάρθρωση. Σκοπό του πιλωτικού προγράμματος ήταν η διευκόλυνση των εργαζομένων στην προσαρμογή τους κατά την περίοδο αναδιαρθρώσεων, με μέτρα τα οποία θα μπορούσαν ε, να καλύψουν ε, την καλύτερη προετοιμασία των εργαζομένων ε, εν ώψη των αλλαγών και ανάλυση και προώθηση καλών πρακτικών. Επί, τη... Επί της αυτής ενημερώσαμε την ε, Επιτροπή σας το 2008 και το 2009 και επίσης δρομολογήσαμε 27 ε, εθνικά σεμινάρια, δηλαδή σε όλα τα κράτη-μέλη, για να μπορέσουμε να αναλύσουμε, να συζητήσουμε για τα μέτρα που αναπτύσσονται στα κράτη-μέλη για να ε, προβλεφθεί και να σύνοδευθεί η αναδιάρθρωση. Συμμετείχαν συνδικάτα, εργοδότες, ε, δημόσιες αρχές και εμπειρογνώμονες. Οι συζητήσεις αυτές βασίστηκαν σε ένα έγγραφο ανάλυσης ε, των εθνικών συστημάτων. Η δεύτερη φάση αφορά την εκπόνηση μιας ε, έκθεσης σύνοψης ε, των ε, διαφόρων εθνικών πρακτικών για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα σε σχέση με τα κοινά στοιχεία, ποιες είναι οι συνθήκες επιτυχίας των καλών πρακτικών τον Απρίλιο του 2009 και τον Ιούνιο του 2010. Στο πλαίσιο της Βελγικής Προεδρίας οργανώσαμε μια μεγάλη διάσκεψη στην οποία συμμετείχαν 500 άτομα για να μπορέσουμε να αναλύσουμε, να παρουσιάσουμε τα συμπεράσματα αυτά και να τα συζητήσουμε. Παρουσία μάλιστα πολλών υπουργών Ένα κοινό στοιχείο υπήρξε, η αναγκαιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο να μπορούμε να έχουμε ένα κοινό πλαίσιο καλών πρακτικών για τη διαχείριση της αναδιάρθρωσης. Και Βάσει αυτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στην ανακοίνωση για την ε, βιομηχανική της πολιτική και στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, πολιτική της για την εσωτερική αγορά, να κάνει διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους για τα ζητήματα αναδιάρθρωσης και βεβαίως Οι εκθέσεις ε, για τα εθνικά συστήματα είναι διαθέσιμες και μόλις ε, παρουσιάσαμε ε, στην Επιτροπή σας τα συμπεράσματα, τα αποτελέσματα, όπως κάναμε και πέρσι, για μια άλλη προσπάθεια την οποία είχε υποστήριξη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η υποστήριξη 18 ε, τομεακών προγραμμάτων που αυτή τη στιγμή ε, όχι μόνο έχουν δρομολογηθεί αλλά αξιολογούνται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Yes, thank you very much. Uh, I think somebody else... Νομίζω ότι και κάποιος άλλος θέλει να πάρει το λόγο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Μάρκο Φέρι και είμαι συντονιστής ε, του Γιούρες και θα απαντήσω στην ερώτηση της ε, κυρίας Σρόντερ για το τι δεν πήγε καλά. Θα προσπαθήσω να σας τα πω σύντομα. Όταν το πιλωτικό πρόγραμμα, πρόγραμμα ε, ξεκίνησε, μας υπευλήθη, για μας ήταν γνωστό, γιατί το 2008-2009 η Επιτροπή σας ε, είχε εκπονήσει μία ε, μελέτη για το θέμα της κινητικότητας και είχατε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει το θέμα των μεταναστών εργαζομένων και των οικογένειών τους. Ε, όταν συζητήσαμε λοιπόν τις κατευθυντήριες γραμμές Γιούρες μαζί με το δίκτυο ε, στη, στα οποία συμμετέχουν κοινωνικοί εταίροι και, τα, και οι δημόσιες αρχές των κρατών μελών. Ε, εμείς προτείναμε αυτήν την ιδέα και έχει συμπεριληφθεί στις κατευθυντήριες γραμμές του Γιούρες. αυτό λοιπόν δεν πήγε καλά. Δεν είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα με την στενή έννοια του όρου. Είναι κάτι το οποίο έχουμε ενσωματώσει ήδη στο Γιούρες ε, που θα το... Ε, αναλάβουμε κατά τα επόμενα δύο χρόνια στο πλαίσιο του Γιούρες, αλλά θα ήθελα να πω δύο ε, πράγματα. Πρώτον, το ποσοστό είναι περίπου 18% το ποσοστό αξιοποίησης των πιστώσεων ε, ανάληψης υποχρεώσεων. Το πρώτο λοιπόν πρόβλημα είναι ότι όταν ρωτήσαμε τα κράτη-μέλη τη ε, δημόσια αρχέ των κρατών μελών αν θέλουν να συμμετέχουν ε, και μέσω μη κυβερνητικών οργανώσεων ε, στην προσπάθεια αυτή, μα είπαν δεν είναι δική μα δουλειά παρά μόνο για συγκεκριμένε περιπτώσει. Οπότε στο τέλο καταλήξαμε με 11 κράτη-μέλη που όντω έχουν πιλωτικά προγράμματα για το θέμα αυτό, αλλά βρισκόμαστε σε μια αρχική φάση και αυτό εξηγεί για ποιο λόγο το ποσοστό είναι τόσο χαμηλό γιατί οι κατευθυντήριες γραμμές ισχύουν για τρία χρόνια, οπότε είπαμε ότι στην αρχή δεν είναι δυνατόν ε, να ε, τα, κάνουμε, τα καταφέρουμε όλα γιατί έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε και γι' αυτό ακριβώς σας εξηγώ γιατί το ποσοστό είναι τόσο χαμηλό. Μετά υπάρχει το θέμα της οικονομικής κρίσης γιατί υπάρχει μεγάλη πίεση ε, για τα κρατημέλη πολλά είναι αυτά που πρέπει να γίνουν και πολλα κρατημέλη κράτη-μέλη μας είπαν δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να κάνουμε κάτι για το θέμα των μεταναστών εργαζομένων γιατί φεύγουν από χώρε στις οποίες δούλευαν. Έχουμε πάρα πολύ καλά παραδείγματα στην Ιρλανδία για παράδειγμα η οποία ε, έχει τέτοιου είδου υπηρεσίες σε μετανάστες εργαζομένου που διαμένουν στην Ιρλανδία. Μέσω μη κυβερνητικών οργανώσεων παρέχουν τι υπηρεσίε αυτέ. και έτσι τους εντάσσουν στην κοινωνία, στην αγορά εργασίας, μέσω εθελοντικής εργασίας κλπ. Κατά την άποψή μου λοιπόν αυτό είναι οι δύο βασικοί λόγοι που μπορούν να εξηγήσουν το χαμηλό ποσοστό απορρόφησης ε, στο πλαίσιο του ε, ε, Και το λέω αυτό γιατί ήταν κυρίως κρατικές υπηρεσίες ε, έβρεσης εργασίας αυτές που συμμετείχαν. Δεν υπήρχαν λοιπόν και πάρα πολλοί, πολλοί πόροι αυτή τη χρονιά, αλλά ελπίζουμε την επόμενη χρονιά, τουλάχιστον αυτή είναι η αίσθηση που είχαμε στις επαφές με τους, ε, με τους εταίρους μας, Ελπίζουμε λοιπόν ότι στο μέλλον θα αποτελέσει ένα καλό παράδειγμα ενσωμάτωσης ε, πιλωτικού προγράμματος ε, στο EURES. Εντάξει, η πρώτη χρονιά δεν ε, έδωσε πολύ καλά αποτελέσματα, ελπίζουμε όμως ε, ότι η επόμενη χρονιά θα πάει καλύτερα και θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις δραστηριότητες αυτές. Γιατί δεν θελήσαμε να εφαρμόσουμε μέσω πιλωτικού προγράμματος. Υπάρχει το θέμα των πόρων, όπως ανέφερε και ο Νικολά, η εφαρμογή ενός προγράμματος ενός εκατομμυρίου ή δέκα εκατομμυρίων ευρώ δημιουργεί κάποιες δυσκολίες. Προτιμούμε να δώσουμε αυτό το χρόνο και τους σπόρους στο Γιούρε. Γιατί? Γιατί είναι ένα δίκτυο που υπάρχει εδώ και 15 χρόνια. Είναι ιδιαίτερο ορατή η δράση του στα κράτη-μέλη. Ε, αυτό αναφέρεται άλλωστε και σε πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρομέτρου και πιστεύουμε λοιπόν ότι στο πλαίσιο του Γιούρες μπορούσαν να αναλυφθούν τέτοιου είδους δραστηριότητες που θα ήταν πιο ορατές στα κράτη-μέλη. Ελπίζω να απάντησα και αν ε, υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις, ευχαρίστω να απαντήσω. Uh, Σας ευχαριστώ, ήταν πολύ χρήσιμα όλα. Ευχαριστούμε πολύ. Η πρόταση για μια τακτική επικοινωνία με την Επιτροπή μας δύο φορές το χρόνο ίσως είναι καλή. Και θα ήθελα βεβαίω να δω ιδιαίτερα για τα συγκεκριμένα πιλωτικά, προγράμματα ε, τις ιδέες σας, για να, τις παρουσιάσεις σας για να βλέπουμε πώς έχουν προχωρήσει. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος χωρίς μικρόφωνο. Η πρόεδρος δεν έχει μικρόφωνο, δεν ακούγεται. presentation by the Commission uh, followed by the rapport. Ολοκληρώνουμε λοιπόν τώρα με τον ε, κύριο Γιάκοπ, ο οποίος θα παρουσιάσει την πρώτη επιτροπή και μετά θα δούμε τον εισηγητή. Κύριε Γιάκοπ, καλό. We've been talking about population Πρόεδρε, έχουμε το θέμα της ε, γύρανσης του πληθυσμού που πλέον, ε, ύστερα από χρόνια που, το, που προειδοποιούσαμε, πραγματοποιείται και γι' αυτό διότι τα παιδιά της εποχής του baby boom έχουν γίνει πια ενήλικες και προχωρούν σιγά σιγά και προς την συνταξιοδότηση. Και έχουμε χαμηλότερη εισρωή εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη. Ενώ ε, αυξάνονται διαρκώς οι αριθμοί των ε, ατόμων με ηλικία των 60 και μάλιστα με ταχύς ρυθμούς. Έτσι λοιπόν τίθεται παρά το ζήτημα και της ε, λειτουργίας των κοινωνιών μας, δηλαδή της απασχόλησης, αλλά και της αλληλεγγύης μεταξύ των ε, διαφορών μερίδων του πληθυσμού. Όμω υπάρχουν ευκαιρίες, υπάρχουν για τους ανθρώπους αυτούς και θέσει απασχόλησης και θελοντικές ε, απασχολήσει και η δυνατότητα της αυτόνομη διαβίωσης χωρίς εξάρτηση δηλαδή εφόσον τους προσφέρουμε το κατάλληλο περιβάλλον. Αυτό είναι που ονομάζουμε ενεργό γύρανση που σημαίνει ταυτόχρονα και αλληλεγγύη μέσα στην κοινωνία μας. Αυτό σημαίνει δράση σε διάφορους πολι... Ε, τομείς πολιτικής και σε διάφορα επίπεδα, τοπικό, περιφερειακό, ε, εθνικό, αλλά και ε, μέσα σε επιχειρήσεις ή σε οργανώσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κεφτεί ένα μερίδιο του καθήκοντος στην υπόθεση αυτή, όπως άλλωστε υπογραμμίζει και, το, και η έκθεση του κ. Μάνολτ. Είδαμε ότι υπάρχουν πολλές ε, μέθοδοι και μέσα, όπως η ανοιχτή μέθοδος συντονισμού και τα διαφορετικά ταμεία με τα προγράμματά τους, αλλά και τα περιφερειακά προγράμματα που μπορούν να προσφέρουν κατάλληλα μέσα για την υποστήριξη στην ενεργογύρανση. η πρόταση για το, την ανακήρυξη του 2011 ως ε, έτους για την ενεργό γύρανση αποτελεί μια ένδειξη από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το πόσο ιδιαίτερη σημασία από στην υπόθεση αυτή και την πρόθεσή της να προσδώσει ορατότητα στις προσπάθειες που αναπτύσσονται σε διάφορα επίπεδα. Έτσι λοιπόν εδώ έχουμε να κάνουμε όχι μόνο με κάποιες ε, ε, εκδηλώσεις που θα έχουν μεγάλη δημοσιότητα μόνο το 2012. Θέλουμε μια ε, δράση συνεχή και ήδη από το 2011 προσκαλούμε τους εμπλεκόμενους φορείς να αναλάβουν αυτούς τους στόχους, έτσι ώστε οι δραστηριότητες αυτές να είναι έτοιμες για το ευρωπαϊκό έτος, για την ενεργογύρανση, αλλά και μετά από το 2012. Πώς θα επιτύχουμε λοιπόν τώρα την αλλαγή προς την ανεργογύρανση. Δεν εξαγοράζεται η δέσμευση στο βαθμό τουλάχιστον που χρειάζεται η ε, κοινωνία μας για να αντιμετωπίσει το ζήτημα της ενεργογύρανσης. Χρειάζεται εμπλοκή εθελοντική, χρειάζεται η βούληση να εμπλακούν οι διάφοροι φορεί στην υπόθεση αυτή. Και έτσι και επειδή είχαμε ευρύτερη ε, υποστηρίξη από την κοινωνία των πολιτών κτλ. θα έχουμε την επιτυχία όπως περιμένουμε. Η επιτυχία του Ευρωπαϊκού Έτους είναι σχεδόν εγγυημένη για μας, όπως τον άλλωστε και η Ευρωπαϊκή ημέρα για την αλληλεγγύη μεταξύ γενεών χωρί την ε, οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το υπογραμμίζω αυτό, διότι εμείς δεν έχουμε στήσει ιδιαίτερο προπολογισμό για το ευρωπαϊκό έτος. Ε, σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε υφιστάμενα κονδύλια. Πολλά ε, κονδύλια είναι διαθέσιμα από διάφορους τομείς και ευρωπαϊκά προγράμματα από την έρευνα, την απασχόληση, την διαβίου μάθηση, ε, που μπορούμε να αξιοποιήσουμε για την ενεργογύρανση. Και έτσι μπορούμε απλώς να δώσουμε την υψηλή προτεραιότητα στις δραστηριότητε για τις ε, ανακοινώσει μας και την επικοινωνιακή μας πολιτική. Ιδιαίτερος προπολογισμός ότι το Ευρωπαϊκό Έντος του άλλους πολύ λίγα θα προσέφερε. Και θα σήμαινε ταυτόχρονα ότι πολύ προσωπικό θα απασχολούνταν στην διαχείριση του ιδιαίτερου αυτού προπολογισμού και έτσι θα μπορούσε να προσφέρει όπω το θέλαμε στι εκδηλώσει του Ευρωπαϊκού Έτου. Και επιτρέψτε μου τώρα να αναφερθώ σε κάποια σημεία που ίσω είναι διαφιλονικούμενα, καταρχά τον τίτλο του Ευρωπαϊκού Έτου. Υπεγράμισα ότι το Ευρωπαϊκό Έτο αναφέρεται στην αλληλεγγύη μεταξύ γενεών. Γιατί λοιπόν δεν αναφέρουμε ακριβώ αυτόν τον τίτλο μέσα στο, στην πρόταση για το Ευρωπαϊκό έτο. Ο τίτλο μα λέει τι πρέπει να γίνει για να διαφυλαχθεί η αλληλεγγύη μεταξύ γενναιών. Είναι σαφής, είναι σύντομος και αυτό είναι ο επικοινωνιακός μας στόχος. Ταυτόχρονα ο τίτλος έχει και την, ε, ε, το πλεονέκτημα ότι δεν παρουσιάζει τον ηλικιωμένο κάποιον ο οποίος χρειάζεται υποστήριξη και βοήθεια ω ένδειξη αλληλεγγύη. Βεβαίω υπάρχουν κάποιοι ηλικιωμένοι οι οποίοι εξαρτώνται από την ελληνική και την υποστήριξη και τη βοήθεια, αλλά υπάρχουν άνθρωποι σε μεγάλη ηλικία οι οποίοι είναι, οι οποίοι είναι δραστήριοι και ικανότατοι. Και ω εκ τούτου θέλουμε να προαγάγουμε τη θετική εικόνα των ηλικιωμένων, των πιο ηλικιωμένων ανθρώπων. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν στην κοινωνία και τον εαυτό του να κοιτάξουν και κάποιον άλλον να κοιτάξουν. Και ακριβώ αυτό θα είναι πιστεύουμε το κύριο μας επιχείρημα και η μεγαλύτερη συμβολή στην αλληλεγγύη μεταξύ γενών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει η πρόεδρος. Ο κύριος Κάσλερ έχει το λόγο ως συγητής. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ την Επιτροπή. Ήταν πολύ καλή η παρουσίαση εδώ για το Ευρωπαϊκό Έτος για το ενεργό γύρανση το 2012 και επέκεινα. Ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Γιάκοπ. Ταυτόχρονα θα ήθελα να ευχαριστώ και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή για την ε, έκθεση της για το θέμα αυτό, για τη σύσταση της μάλλον. Θα είναι πολύ χρήσιμη οι προτάσεις της για το Κοινοβούλιο στην ε, παρούσα στιγμή. Είναι βέβαια θέμα επικαιρότητα όχι μόνο στι Βρυξέλλες, η ενεργός γυράνση, αλλά και παντού στην Ευρώπη. Είναι σαφές αυτό αν δούμε τις διαρκείς εξελίξεις, ε, τη δημογραφική εξέλιξη στην Ευρώπη. Τι συνέπειες που αυτή θα έχει και στην παροχή των υπηρεσιών, της ταξιδιωτικά συστήματα και το καθεξής. Και γι' αυτό νομίζω ότι αυτή η πρωτοβουλία που σημαίνει ταυτόχρονα και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης, καλύτερες συνθήκες απασχόλησης για τους πιο ηλικιωμένους στην Ευρώπη, ε, αποτελεί μια πολύ καλή ε, πρόταση και ταυτόχρονα καλούμεθα να απαντήσουμε στο ερώτημα πώς μπορούν οι πιο ηλικιωμένοι να προσφέρουν και στο χώρο εργασίας και πώς μπορεί να προαχθεί η παρουσία και η συμβολή τους αυτή. Εδώ, ιδιαίτερα με την αρχή της επικουρικότητας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ρόλο συντονιστικό και ταυτόχρονα καλούνται οι τοπικές, περιφερειακές αλλά και εθνικές αρχές σε ε, σύμπραξη με την κοινωνία των πολιτών, όπως επισήμανε και ο κύριος Γιάκοπ, τους κοινωνικούς εταίρους δηλαδή, να αναπτύξουν πρωτοβουλίες και να τις εφαρμόσουν το 2012. Εγώ ως εισηγητής υποστηρίζω την ε, πρόταση, την έμφαση που δίνεται στην ε, κοινωνική αλληλεγγύη μετά την Ευρωπαϊκή Χρονιά για την καταπολέμηση της ένδυας. Το 2011 θα είναι το Ευρωπαϊκό έτος για την εθελοντική απασχόληση και το 2012 όπως είπατε και εσείς ο ίδιος και Γιάκο μπορεί να έχει να προκαλέσει κάποιες αντιδράσεις προς τον τίτλο του. Ναι, το, ο τίτλος του έτους θα έχει ιδιαίτερη σημασία και πρέπει να το συζητήσουμε όταν έρθει η ώρα να δούμε εάν η έννοια της γενεάς πρέπει να ενσωματωθεί μέσα στον τίτλο και αν πρέπει με κάποιο τρόπο να συνδέσουμε τις, δύο, τις διάφορες γενναίες μεταξύ τους. Αυτό είναι το ένα που πρέπει να συζητήσουμε. Και δεύτερον, χωρίς όμως να το θεωρώ κεντρικό σημείο της συζήτησης, το ζήτημα της γραμμής του προπολογισμού, που είπατε ότι δεν θα, κατα... δεν θα ζητήσετε και αιτιολογήσετε και την επιλογή σας. Ασφαλώς όμως θα προκαλέσει αρκετά ερωτηματικά αυτή η επιλογή γιατί ευρωπαϊκό έτος χωρίς κονδύλια τι μπορεί να προτείνει. Είπατε ότι έχετε και τις δομές, έχετε τις γενικές διευθύνσεις, αναφέρατε και ο ίδιος. Είπατε ότι θα αναλάβουν δραστηριότητα στον τομέα αυτών. Έχω όμως μια σημαντική ερώτηση εν προκειμένου. Εάν ένα ευρωπαϊκό έτος μπορεί να προχωρήσει χωρίς δικό του προϋπολογισμό. Πρόκειται για μια ερώτηση την οποία ασφαλώ θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε. Και περιμένω μια εντατική συζήτηση, όχι μόνο για το, και τον αλλά και για τον προπολογισμό, αλλά και γενικότερα, διότι με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με τη βάση ε, πρόταση της, ε, της, τη σχετική με τα κοινωνικά ζητήματα, έχουμε νομίζω μια καλή βάση για συζήτηση. Είμαστε εξοπλισμένοι στην υπόθεση αυτήν και ως εκ τούτου μπορούμε να προχωρήσουμε και με τον σκιώδη συγκητή και τους συγκητές από τις... Ε, με τον τον κύριο αλλά και με τους σκιώδη συγκητές γιατί έχουμε δύο ακόμη αρμόδιες ε, για ε, γνωμοδότηση επιτροπές, ε, την οικονομική και την πολιτισμού, που νομίζω ότι μπορούμε να ε, εμπλέξουμε στην όλη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Σας... Σας ευχαριστώ πολύ. Έχω και εγώ μια-δυο ερωτήσεις. Όπως και εσείς είπατε, πρέπει να δούμε το θέμα αυτό ως ευκαιρία. Πολύ συχνά όταν μιλάμε για την κύρανση και τον κυράσκοντα πληθυσμό και λέμε ότι πρέπει να ασχοληθούμε και με τους νεότερους. Πολλοί πιστεύουν ότι είναι αρνητική γύρανση του πληθυσμού, Είναι αρνητικό φαινόμενο. Όμως το θέμα είναι να λάβουμε υπόψη το τι γίνεται με τους ηλικιωμένους ανθρώπους. Να δούμε αυτήν την διάσταση. Τα κάτι μελη καμιά φορά αντιμετωπίζουν το θέμα αυτό σαν ορολογιακή βόμβα και οι εφημερίδες έτσι το προβάλλουν με πολύ αρνητικές αποχρώσεις. Λοιπόν πρέπει να δούμε τα αποτελέσματα όπως λέτε. Έχουμε τόσα ευρωπαϊκά έτη για τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, για τόσα πολλά θέματα. Ε, είχα ανέκαθεν την αίσθηση ότι όλες οι συνεδριάσεις, ε, τα συνέδρια που διοργανώνται στα κράτη-μέλη είναι πολύ ως ευκαιρίες για να μιλάει ο καθένας με αφορμή το κάθε έτος και το θέμα στο οποίο είναι αφιερωμένο, αλλά στο τέλος δεν αναλαμβάνεται δράση, δεν προχωρούν ε, οι στόχοι και οι προτεραιότητές μας. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα για αυτό που μας είπατε και ξέρω ότι το Κοινοβούλιο θέλει να δείτε τα θετικά αποτελέσματα από αυτό το ευρωπαϊκό έτος. Ένα από τα πιθανά αποτελέσματα, και αυτό μας απασχολεί ιδιαίτερος, όπως έγινε με το έτος για τους ανθρώπους με αναπηρίες, ήταν να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε τέτοιο είδο νομοθεσία που θα επιτρέψει να αναλυθεί δράση για την προστασία των ανθρώπων με αναπηρίες. Αυτό βεβαίω απαιτούσε μια οριζόντια οδηγία που αυτή τη στιγμή που ξέρουμε στο Συμβούλιο. Αλλά πόσο σημαντικό θεωρείτε εσείς ότι είναι να λάβουμε αυτό το χαρτοφυλάκιο από το Συμβούλιο πριν το 2012 ελπίζω Πρέπει να κινηθούμε και προς αυτή την κατεύθυνση, διότι μιλάμε για δραστηριοποίηση. βεβαίω υπάρχει η οδηγία περί απασχόλησης το 2000 κατά της ε, διακριτική μεταχείριση και στην απασχόληση στην εργασία. Ξέρω ότι από κάποια μέλη εφαρμόζεται, υλοποιείται, αλλά όσοι δεν έχουν πρόσβαση σαν τις οδηγίες αυτής, τελικά δείχνουν ότι η οδηγία αυτή καθίσταται κοινή νοήματος. Υπάρχει οδηγία για τη διακριτική μεταχείριση, για την πρόσβαση στα αγαθάκια και τι για του ανθρώπου με αναπηρίε, σε σχέση με τι θρησκευτικέ του πεπιθήσει και του σεξουαλικό του προσανατολισμό. Ε, νομίζω λοιπόν ότι υπάρχουν εδώ κάποια προσκόμματα, αλλά πώ μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό το ευρωπαϊκό έτο, πιστεύετε εσεί, ασκώντα πίεση στα κράτη-μέλη. Δεν είναι μόνο ένα αυτό που παρακολεί τη διαδικασία κατά την άποψή μου. Υπάρχει ένα το οποίο ανθίσταται περισσότερο από τους υπόλοιπους, αλλά και άλλοι κρύβονται πίσω του. Το έχουν βάλει μπροστά και αποφεύγουν. Πώς μπορούμε λοιπόν να αξιοποιήσουμε το έτος αυτό, ώστε να έχουμε ένα πραγματικά θετικό αποτέλεσμα. Να την αποσπάσουμε πλέον αυτή την οδηγία, μια διαπαντό. Εδώ κάνουμε εκστρατείες εδώ και 11 χρόνια για να περάσει αυτό. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει αυτό το θετικό αποτέλεσμα. Ότι θα γίνει πραγματικότητα. Εάν μπορούσατε λοιπόν να επεκταθείτε και σε αυτό και σε άλλα πιθανά θετικά αποτελέσματα που πιστεύω ότι μπορούμε να επιτύχουμε. Πού βρίσκεται το Συμβούλιο για τα θέματα αυτά. Για τον προπολογισμό. Και εγώ το είδα και σκέφτηκα ότι είναι περίεργο αυτό με τη δημοσιονομική γραμμή. Αλλά και από όσα είπατε προκύπτει το εξή ερώτημα. Πιστεύετε ότι οι πόροι, τα κονδύλια εντοπίστηκαν από υπάρχοντες προπολογισμούς. Χρήσιμο θα ήταν για τις μελλοντικέ μας συζητήσεις της Επιτροπής να ξέρουμε τη δική σας άποψη για το πού θα, από την πηγή από την οποία θα προέρχονται αναλυτικά τα κονδύλια. Ακόμη και γραπτό, αν γίνεται να μα το στείλετε, ώστε όλοι στην Επιτροπή μα να έχουν αυτά τα πιστήρια στα χέρια του, αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία. Πολλοί είναι αυτοί που πιέζουν για μια συγκεκριμένη δημοσιονομική γραμμή και θέλουμε να την πάρουμε. Είναι σημαντικό λοιπόν να ξέρουμε από πού αποδίδονται αυτά τα κονδύλια. Εάν τα ευρωπαϊκά έτη επιτρέπουν να τεθούν σε δράση, να σχεδιαστούν μάλλον σε δραστηριότητε που θέλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω αν άλλοι βουλευτέ θέλουν τον λόγο. Παρακαλώ. Euh, Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Έχετε δίκιο να λέτε ότι είναι σημαντικό κάποιο ευρωπαϊκό έτος και για το συγκεκριμένο θέμα ένα τέτοιο έτος θα πρέπει να αποφύγουμε την περίπτωση των ευρωπαϊκών ετών με πολύ ωραία λόγια αλλά χωρί κανένα νόημα. Εδώ χρειαζόμαστε συγκεκριμένε δράσει. Πριν το τέλο του έτου θέλουμε να θεσπιστεί μια στρατηγική που να οδηγήσει σε συγκεκριμένα εργαλεία. Ένα από τα βασικά προβλήματα, και το είδαμε κατά το έτο πολέμηση τη ένδυα, είναι ότι όλο και περισσότερο οι ηλικιωμένοι γίνονται και φτωχότεροι. Θέλω να θέσω λοιπόν το εξή ερώτημα. Η ιδέα τη οδηγία πλαισίου για το ελάχιστο εισόδημα θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτηση. Αυτό είναι ένα πρώτο στοιχείο. Έπειτα, δίκαιο έχετε όταν λέτε ότι θα πρέπει το έτος αυτό να το δούμε από την ε, σκοπιά την, της θετικής προσέγγισης. Ας βασιστούμε όμως πρώτα απ' όλα στην πείρα των ε, ηλικιωμένων πολιτών, ώστε να μπορέσουν να περάσουν στην κατάρτιση, την επαγγελματική κατάρτιση. Ακριβώς δηλαδή να φροντίσουμε οι νέοι που φτάνουν στις επιχειρήσεις να καταρτίζονται, να εκπαιδεύονται από τους ηλικιωμένους με τις γνώσεις και την τεχνογνωσία τους. Αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο. Και το τρίτο είναι ότι δεν μπορούμε να ξαναδημιουργήσουμε μια κοινωνία αλληλεγγύης εάν δεν επιμείνουμε στην αλληλεγγύη μεταξύ των διαφορετικών γενεών. Εδώ δεν μπορούμε να φέρνουμε σε αντιπαράθεση τους νέους με τους ηλικιωμένους. Πρέπει να συνεπάρξουν ειρηνικά. Αυτό νομίζω ότι είναι ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της δικής σας της δουλειάς και κατά συνέπεια ελπίζω ότι θα αξιοποιήσετε αυτές τις λίγες ιδέες που σας εξέθεσα και μάλιστα σύντομα. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστούμε. Η κυρία Μπλενκεβιτσιούτε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάληψη αυτή τη πρωτοβουλία και την παρουσίαση που μας έκανε για το Ευρωπαϊκό Έτος τη ενεργού γύρανση. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, γιατί και ταχύτατα ο πληθυσμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι αλήθεια ότι θα πρέπει από το φαινόμενο αυτό να αναζητήσουμε και τι θετικέ του πτυχέ. Πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε αλληλέγγυοι με του ηλικιωμένου πολίτε τους μεγαλύτερου από εμά. Όμως δεν μπορώ να συμφωνήσω απολύτω και με μια πρωτοβουλία της Επιτροπής ε, που οδεύει στην εξή κατεύθυνση. Δεν μιλούμε αρκετά για την απασχόληση των ηλικιωμένων, για τη δυνατότητα που έχουν να βρουν δουλειά στην αγορά εργασία Αυτό είναι μείζονο σημασία. Ιδίω όταν πρόκειται για κάτι που σχολιάζεται και σε μια πράσινη βίβλο. Δηλαδή, ε, ε, όλοι θα δουλεύουμε περισσότερο χρόνια στο μέλλον. Η Επιτροπή δεν μας έχει υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για την απασχόληση των ε, ηλικιωμένων πολιτών. Εάν δεν συμβεί λοιπόν κάτι τέτοιο, δεν μπορούμε να συζητούμε για ένα θέμα τόσο μεγάλη σημασία. Όπως είναι η παράταση του χρόνου εργασίας πριν τη συνταξιδότηση. Στα πλαίσια λοιπόν της ενεργούς γύρανσης δεν μπορούμε να μείνουμε μόνο στην απασχόληση, ούτως ή άλλως θα πρέπει να διασφαλίσουμε τις ε, κατάλληλες υποδομές, να παρέχονται οι κατάλληλες υπηρεσίες προς τους ηλικιωμένους, το κατάλληλο υγειονομικό σύστημα και η περίθαλψη. Όλα αυτά είναι απαραίτητα αν θέλουμε οι ηλικιωμένοι να παραμείνουν ενεργοί για περισσότερο χρονικό διάστημα. Για το περιβάλλον και την προσαρμογή του επίση πρέπει να μιλήσουμε βάσει των αναγκών των ηλικιωμένων, αν θέλουμε να παραμείνουν δραστήρια μέλη τη κοινωνία. Η συμμετοχή των ε, ηλικιωμένων πολιτών σε μη κυβερνητικέ οργανώσει και αυτό πρέπει να προαχθεί. Δεν ξέρω αν το Ευρωπαϊκό Έτο τη Ανεργού Κυρία θα δώσει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Λένε πολλοί ότι όχι, όχι, δεν χρειάζεται προπολογισμό γιατί έχουμε άλλα προγράμματα, άλλε προτάσει. Δεν έχουμε αρκετά χρήματα, αρκετού πόρου. Όμως για να έχουμε αποτελέσματα απαιτείται προπολογισμό. Χρειάζεται οδηγία κατά της διακριτικής μεταχείρισης. Χρειάζεται άλλη οδηγία για την καταπολέμηση της διακριτικής μεταχείρισης κατά των ε, ηλικιωμένων. Όλα αυτά θα επιτρέψουν να συντονίσουμε καλύτερα τις δραστηριότητές μας. Δραστηριότητες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων για να μην καταλήξουμε σε αντιφάσκοντα αποτελέσματα το Ευρωπαϊκό Έτος Καταπολέμησης της Ένδειας, όπως ξέρουμε, δεν έδωσε συγκεκριμένα αποτελέσματα ακόμη. Κάποια κράτη, συγκεκριμένα κράτη, ε, αύξησαν τον αριθμό των ε, πολιτών που έχουν προβλήματα φτώχειας, αντί να το μειώσουν. Λοιπόν αυξάνεται ο αριθμό των ανθρώπων που έχουν ανάγκη από βοήθεια από την κοινωνία, από κοινωνική βοήθεια. Δεν έχουν αρκετά μέσα για να εξασφαλίσουν τη διαβίωσή του. Αυτά. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, ευχαριστώ. Έχετε να προσθέσετε κάτι κύριε Κάσλα. Δίνω το λόγο κατευθείαν στην Επιτροπή. Έχετε κάποιο σχόλιο να κάνετε. Also ich möchte zwei Dinge noch... Σε ένα-δύο πράγματα θέλω να αναφερθώ. Για τον προπολογισμό ήδη αναφέρθηκε ότι θα πρέπει να συζητηθεί η επιλογή και αν θέλουμε να ανακηρύξουμε ένα ευρωπαϊκό έτος για την ενεργογύρανση καλό θα είναι να μην περιοριστούμε μόνο στην απλή δημοσίευση μιας σειράς ε, προσπέκτους και γράφων. Ήθελα επίσης να επισημάνω ότι ε, δίνεται με το ευρωπαϊκό Έτο μια ευκαιρία να συζητήσουμε πράγματα τα οποία δεν συζητούνται εν γέννη ή να τα συζητήσουμε πολύ πιο εντατικά. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο θεωρώ ότι είναι σημαντικό να έχουμε το ευρωπαϊκό έτος για, το ενεργό, για την ενεργό γύρανση, έστω και αν δεν δούμε άμεσα τα αποτελέσματα, γιατί βλέπουμε ότι ούτω ή άλλω οι δομέ, οι ευρωπαϊκέ, οι κοινωνικέ δομέ θα αλλάξουν σταδιακά και έτσι θα δούμε και να εμφανίζονται οι πιο ηλικιωμένοι ε, που είναι διατεθειμένοι να στρατευτούν, να δραστηριοποιηθούν σε διάφορες περιπτώσεις, σε υπηρεσίες μέσα στην οικογένειά τους, να προσφέρουν σε θελοντικό, φιλανθρωπικό έργο, σε φροντίδα για κάποιους άλλους. Όλα αυτά λοιπόν λαμβανόμενα υπόψη μας οδηγούν στο συμπερασμό ότι είναι σημαντικό και για όποιον θέλει να κάνει αυτή τη δουλειά, που θέλει να δραστηριοποιηθεί ως ηλικιωμένος, να έχει την αναγνώριση του ευρωπαϊκού έτους. Επομένως το ζήτημα δεν, είναι, δεν εξαντλείται μόνο στην απασχόληση, αλλά στο πόσο μπορεί ο ηλικιωμένος, ο πιο ηλικιωμένος, να προσφέρει στην κοινωνία και σε αυτήν ακριβώς την προσφορά θέλουμε να εξασφαλίσουμε αναγνώριση μέσω του Ευρωπαϊκού Έτους. Με αποτελέσματα τα οποία ξέρουμε δεν θα πραγματοποιηθούν από τη μία μέρα στην άλλη. Αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε τη σχετική προσπάθεια για να, προσ... για να βελτιωθεί η πρόταση, την οποία ήδη όμως θεωρώ αρκετά καλή. Ευχαριστώ. Uh, thank you. I'm back. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ιδιαίτερω όλους τους βουλευτές που έλαβαν το λόγο για τη στήριξη που έδωσαν σε αυτό το εγχείρημα. Είναι πολύ ενθαρρυντικό. Να κάνω μια γενική παρατήρηση. Η... Τα ευρωπαϊκά έτη είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, διότι το θέμα της ενεργού γερανσής δεν είναι κάτι που μπορούμε να το δούμε από το ευρωπαϊκό επίπεδο προς τα κάτω μόνον. Πρέπει να αναλυθούν πολλές δράσεις και σε επίπεδο κρατών μελών, σε επίπεδο τοπικών αρχών, εταιριών και το καθεξής. Αυτό που μπορούμε να προσφέρουμε είναι ένα πλαίσιο. Ένα πλαίσιο το οποίο να ευαισθητοποιήσει και να ασκήσει κάποια πίεση σε όλα αυτά τα διαφορετικά επίπεδα, ώστε να αναλυθεί η δράση. Η πίεση αυτή θα πρέπει να ασκηθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μιλήσατε, Πρόεδρε, για μια οδηγία. Βεβαίω, το να οργανωθεί ένα ευρωπαϊκό έτο ε, προβάλλει και ενημερώνει καλύτερα για τα προβλήματα διακριτική μεταχείριση. Αυτό το είδο λοιπόν η προβολή θα μα διευκολύνει. Θα επιτρέψει να έχουμε επικοδομητικότερη συζήτηση στο ευρωπαϊκό επίπεδο για τα θέματα αυτά. Θετικά αποτελέσματα τώρα. Πρέπει να επιτευχθούν τέτοια αποτελέσματα σε όλα τα επίπεδα. Σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό, εγώ θα ανέμενα τέτοια θετικά αποτελέσματα και επειδή βλέπω ποια είναι η φιλοσοφία των συναδέλφων σε διάφορες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γνωρίζουν εκείνοι τι δυνατότητες έχουν μέσω των προγραμμάτων και των πολιτικών και των πολιτικών πρωτοβουλειών που οργανώνονται για να συμβάλλουν στους στόχους της ενεργού γύρανσης, ε, είναι ένα θέμα που έχει γίνει θέμα προτεραιότητα σε πολλέ υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με πολλού συναδέλφου. Ένδοεπηρεσιακώ. Βλέπουμε λοιπόν να υπάρχει ισχυρή κινητοποίηση ω προ την ενεργογύρανση. Και έρχομαι τώρα στο θέμα τη δημοσιονομική γραμμή. Ρωτήσατε εάν μπορούμε να έχουμε μια λεπτομερή ανάλυση των κονδυλίων που μπορούμε να αποσπάσουμε, να, να εκταμιεύσουμε για να χρηματοδοτήσουμε τα ζητήματα τη ενεργού γύρανση. Το, έχει, το έχουν συζητήσει αυτό και οι υπουργοί στο Συμβούλιο των Κοινωνικών Υποθέσεων και καλωσορίσαμε τα συμπεράσματά του. Και η πρώτη συνάντηση με του εκπροσώπου των κρατών μελών ε, θα γίνει σύντομα, ώστε να δούμε ποιε είναι οι δικέ του προσδοκίε και να μπορέσουμε να συντονίσουμε του δικού μα πόρου με τι ανάγκε που υπάρχουν, ώστε να δούμε κατά πόσον τα κονδύλια αυτά μπορούν να κατευθυνθούν προς τα κάτι μέλη. The... Επίσης, έγιναν αναφορές στις ανάγκες που πρέπει να αντιμετωπιστούν στα θέματα της ενεργού γύρανσης, όπως ο ρόλος των ηλικιωμένων στην επαγγελματική κατάρτιση. Εδώ νομίζω ότι έχουμε ένα σαφές παράδειγμα του τι θα μπορούσαμε να προάγουμε. τι πρωτοβουλίε δηλαδή μπορούμε να οργανώσουμε στο ευρωπαϊκό έτο. Ήδη το 2011 έχουμε κανονίσει συναντήσει με συνομιλητέ και εταίρου σε διαφορετικά επίπεδα για να αρχίσουν να σκέφτονται τι μπορούν να κάνουν ώστε να συμβάλλουν στην ενεργοκύρανση. Οι δεσμεύσει αυτέ θα δημοσιοποιηθούν. Θα τι βάλουμε σε έναν ιστότοπο ώστε όλοι να μπορούν να τι δουν. Θα βλέπουν τι σχεδιάζει ο κάθε ένα από του διαφορετικού φορεί και συνομιλητέ μα. Οι πρωτοβουλίε εκπαίδευση είναι κάτι που επιτρέπει στου να περάσουν τις γνώσεις τους στους νεότερους. Συμφωνώ απολύτως. Υπάρχει ανάγκη να βελτιωθούν οι υποδομέ υπηρεσιών για του ηλικιωμένου, για να δημιουργηθεί ένα γιέστερο περιβάλλον. Βεβαίω αυτό είναι μέρο ε, του προγράμματο για την ε, ενεργογύρανση, κυρίω για την βελτίωση τη διαβίωση των ηλικιωμένων. again. Και μια τελευταία παρατήρηση για την ελληνική μεταξύ των διαφορετικών γενεών. Ναι, το έτος αυτό αφορά και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενναίων. Όμως θέλουμε να προωθήσουμε τα πράγματα αυτά από μια διαφορετική προοπτική από τη συνηθισμένη. Δηλαδή, να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες των ηλικιωμένων, κινητοποιώντας αυτούς τους ίδιους, ώστε να συμβάλλουν στην κοινωνία. Αυτό θεωρούμε ότι είναι ακόμη πιο σημαντικό, ώστε να μην τους αντιλαμβάνονται άλλοι ως βάρος δεν είναι βάρος. Μπορούν πολλά να δώσουν και πρέπει να τους αφήσουμε. Πρέπει να δημιουργήσουμε συνθήκες τέτοιες ώστε να μπορέσουν και εκείνοι να συνεισφέρουν. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Όταν θα έχετε ολοκληρώσει την συγκέντρωση των γραμμών του προπολογισμού από τους διάφορους προπολογισμού, θα θέλαμε να μας αποστείλετε τον κατάλογο το συντομότερο δυνατόν. Γνωρίζετε το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας αυτής, γιατί είναι ένα από τα βασικότερα ε, ζητήματα που μας ενδιαφέρουν. Δεν, υπάρχουν, δεν υπάρχει γραμμή προπολογισμού. Ίσως θα μπορούσατε να μας πείτε ότι θα υπάρξει κάτι, να γνωρίζουμε πάση περιπτώσει από πού θα προέλθουν τα κονδύλια. Προβλέπουμε να γίνει κατά τέτοιο στο επόμενο δεκαπενθήμερο και θα το συζητήσουμε σε μία συνεδρίαση που έχουμε προγραμματίσει με τα κράτη-μέλη στις 30 Νοεμβρίου. Εντάξει, λέει η Πρόεδρος, θα ήταν χρήσιμο να ενημερώσετε και την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Ζητημάτων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι για την παρουσίασή σας. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η βιομηχανική πολιτική σε μια ε, εποχή παγκοσμιοποίησης, σε εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης. Δίνω το λόγο στον εισηγητή. Τον κύριο Λούτβιξον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι συντάκτης γνωμοδότησης για το θέμα αυτό και για όσους δεν είχαν το χρόνο να διαβάσουν την γνωμοδότησή ε, μου. Θα ήθελα να πω καταρχάς ότι χρειαζόμαστε μία ισχυρή ανταγωνιστική βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει κοινωνική συνοχή και επίση να εξασφαλίσουμε ότι οι ευρωπαϊκές θέσεις απασχόλησης είναι καλές θέσεις απασχόλησης και να μπορούμε επίσης να καταπολεμήσουμε και την ανεργία. Η αναδιάρθρωση λόγω της ε, παγκοσμιοποίησης πρέπει να γίνει στο πλαίσιο ενός κοινωνικού διαλόγου. Τώρα, η μετάβαση στην ε, πράσινη οικονομία πρέπει να γίνει με δίκαιους όρους. Πρέπει να υπάρξει καινοτομία, επενδύσεις και πρέπει να δημιουργήσουμε νέες πιο πράσινες θέσεις απασχόλησης και στον τομέα της βιομηχανίας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επενδύσουμε στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων ώστε να μπορούν οι πολίτες να διατηρήσουν τις ε, θέσεις απασχόλησής τους ακόμη και μετά από την αναδιάρθρωση και επίσης να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις μελλοντικέ ανάγκες της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Όσον αφορά τώρα το διασυνοριακό πλαίσιο για τι συλλογικέ διαπραγματεύσει και τι σχετικέ εργασίε Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρά το γεγονό ότι είναι εκτό ε, αρμοδιότητα Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν, υπάρχουν άλλοι τομεί για του οποίου το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο. Για παράδειγμα, ε, οι όροι πρόσληψη, η συνεχιζόμενη κατάρτιση ή το πώ ε, οργανώνεται η εργασία. Εγώ πραγματικά Αναμένω εναγωνίω τα σχόλια των συναδέλφων και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 15 Νοεμβρίου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανείς άλλο συνάδελφος να πάρει το λόγο σε σχέση με την ε, βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίηση. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και θέλω να ευχαριστώ τον ε, εισηγητή για τις προτάσεις του. Ήδη φαίνεται ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ των υπόψεων του εισηγητού και της δικής μου ομάδας. Τον ε, ευχαριστώ λοιπόν και τον υποστηρίζω στην καιροτομία στους νέους τομείς τεχνολογίας. Πρέπει να προχωρήσουμε κατά τρόπο μη ε, επιλεκτικό και να αφήσουμε την επιλογή στην ε, προώθηση συγκεκριμένων τεχνολογιών στην αγορά. Πρέπει να διευκολύνουμε την αποδοχή και κατανόηση από τον πολίτη της τεχνολογίας. Ιδιαίτερα δε σημαντικός παράγων και, και εκ των όνων κάνευ όρος είναι η κατάρτιση των πολιτών, έτσι ώστε να έχουμε ένα εργατικό δυναμικό με τις κατάλληλες δεξιότητες και η ανάπτυξη των σχετικών θέσεων εργασίας. Όταν λοιπόν μιλούμε για ε, εκβιομηχάνηση στην Ευρώπη, για καλύτερα διαφύλαξη των θέσεων εργασίας στο βιομηχανικό τομέα στην Ευρώπη, τέτοιου είδους θέσεις είναι απαραίτητες. Τέτοιου είδους θέσεις ψηλή τεχνολογία τεχνολογίας αιχμή, μπορούν να αποτελέσουν το 37% τη βιομηχανική δραστηριότητα στην Ευρώπη. Ενώ βλέπουμε ταυτόχρονα ότι ένα υπουργό μιλάει στον Ηνωμένο Βασίλειο για 6 μόνο τη 100 κάλυψη ε, τη βιομηχανική δραστηριότητα από τέτοιου είδου θέσει αυτή τη στιγμή. Ο στόχο μα θα πρέπει να είναι λοιπόν να τι πολλαπλασιάσουμε. Έναντι των μεγάλων ανταγωνιστών έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών κυρίως υποβαθμιζόμαστε εφόσον δεν έχουμε τέτοιου είδου εργατικό δυναμικό υψηλή κατάρτισης και τεχνολογίας σε έναν χώρο μόνο παροχής υπηρεσιών και βέβαια σε πολύ ψηστά ε, ποσοστά ανεργίας το οποία καλούμεθα να διαχειριστούμε. Έχουμε θέματα λοιπόν που είναι και της Επιτροπής Απασχόλησης και της Επιτροπής για την Ιστορική Αγορά που εγώ έχω την ε, ε, εισήγηση αναλάβει, την έκθεση αναλάβει ε, και πρέπει να επιδιώξουμε, να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας στον χώρο αυτών και πράσινο να είναι ο Εγώ δεν έχω καμιά αντίρρηση πρόβλημα με τέτοιου είδου επιλογέ πράσινε, διότι βλέπουμε όχι μόνο στη Γερμανία αλλά και σε όλη την Ευρώπη ότι η πράσινη ιδεολογία και πολιτική προάγει νέε τεχνολογίε ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια και τι σχετικέ τεχνολογίε του, οι οποίε μπορούν να σημάνουν και περισσότερη απασχόληση για τους πολίτες μας. Εκεί λοιπόν θα πρέπει ίσως να διατυπώσουμε τις ε, απαιτήσει μα έτσι ώστε στο μέλλον η Ευρώπη να παραμείνει χώρος και παραγωγή να μην υποβαθμιστεί, να αναβαθμιστεί μάλλον και να μην χαθούν οι θέσει εργασία. Να υπάρξουν νέε θέσει εργασία στις καινοτόμε βιομηχανίε, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε καλύτερε ευκαιρίες για κάθε Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ κύριο Σάνγκλη. Πρόεδρε ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ ξεκινώντας να πω ότι το σχέδιο του εισηγητή νομίζω ότι συμπεριλαμβάνει τα σημαντικότερα σημεία. Ο ή πρόκειται για γνωμοδότηση. Οπότε δεν έχουμε και απεριόριστο χώρο για να επεκταθούμε στην ανάλυση όλων των ανησυχιών μας. Έχω την εντύπωση ότι σε γενικές γραμμές είναι σημαντικό να ξέρουμε τι βιομηχανίες θα έχουμε στο μέλλον στην Ευρώπη. Αυτό έχει να κάνει και με το τι συμβαίνει με το βιομηχανικό μας χώρο και πώς εξελίσσεται στο Λουξεμβούργο. Η βιομηχανία εκπροσωπεί το 19% του εγχώριου προϊόντος. Ε, κάτι ανάλογο φαίνεται να συμβαίνει και στα υπόλοιπα κράτη και αυτό βεβαίως έχει τις επιπτώσεις του στην απασχόληση. Η βιομηχανία Λοιπόν, πρέπει να δούμε αν θα μας οδηγήσει σε ένα φαινόμενο αποβιομηχανοποίησης της Ευρώπης. Δηλαδή, σίγουρα η βιομηχανία δίνει κάποια απασχόληση, θέσεις απασχόληση σε ανθρώπους που τη χρειάζονται, ε, αλλά πάνω απ' όλα σε αυτούς που δεν έχουν τα ψηλότερα προσόντα. Πρέπει λοιπόν να είμαστε αποφασιστικοί ω προ την ευρωπαϊκή δέσμευση για τη στήριξη τη βιομηχανία στο μέλλον. Να είμαστε προσεκτικοί ω προ το ότι ενώ συνεχίζουμε να κατηγορούμε και να κρίνουμε την Κίνα που στα περιβαλλοντικά και περισσότερο στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών βρίσκεται στο, μεταξύ των τελευταίων που κάνουν κάτι. Όμως φέτος η Κίνα επένδυσε περισσότερο στις πράσινες τεχνολογίες από οποιονδήποτε άλλο στον κόσμο. Και αυτή είναι μια παγιωμένη κατάσταση που μάλλον θα συνεχιστεί. Η Κίνα δημιουργεί θέσει εργασία σε αυτό το τομέα, ενώ η Ευρώπη μένει πίσω. Και μετά τι ε, προτάσει του ε, Επιτρόπου που είναι επιφορτισμένο με τα θέματα ενέργεια, μα μίλησε για ευρωπαϊκέ επενδύσει από τώρα στο 2020 για να τελειοποιήσουμε το ενεργειακό μα σύστημα. Αυτό αφορά άμεσα την βιομηχανία, άμεσα τις, αποτελεσμα... τις της ε, εργασίας στον τομέα της τεχνολογίας και της βιομηχανίας. Είναι όλα αυτά ιδέες που θα πρέπει να τις ε, μελετήσουμε. Πάντως, βρισκόμαστε ακόμα στα προκατακτικά στάδια. Εγώ πιστεύω ότι πέρα από κάποιες ωραίες εκφράσεις επιπλέον δεν θα έχουμε και πάρα πολλά να πούμε τόσο άμεσα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Ντελή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας για, το, για τη δουλειά του και να σταθώ σε αρκετά στοιχεία. Βρισκόμαστε σε μια ιστορική στιγμή αλλαγής απέναντί μας έχουμε την κατεξοχήν πρόκληση, την κλιματική πρόκληση. Δεν είμαι εγώ που το λέω, το λένε όλοι και είναι κατεπήγον. Η κλιματική λοιπόν πρόκληση οδηγεί και σε κοινωνικές δυσκολίες. Βεβαίως θα χρειαστούν μετατροπές και περάσματα σε νέες μορφές επαγγελματικές. Αυτές οι μεταβολές, αυτές οι Μετακινήσεις θα πρέπει να γίνουν με ενθάρρυνση των εργαζομένων από την επαγγελματική κατάρτιση να αναζητήσουν νέα θέση εργασίας Νομίζω ότι η ασφάλεια εδώ είναι ένας παράγων που θα πρέπει να μας απασχολήσει. πώς θα οργανώσουμε το μεταφατικό εισόδημα των ανθρώπων αυτών, αυτοί που αλλάζουν επάγγελμα. Πώ θα εξασφαλίζουν τη διαβίωσή του κατά την περίοδο της μετάβαση. Αυτό είναι ένα πρώτο στοιχείο. Πρέπει λοιπόν να θυμίσουμε ότι η επαγγελματική κατάρτιση είναι σημαντική, ότι το μεταβατικό εισόδημα χρειάζεται και επίση η κατάρτιση πρέπει να είναι μια κατάρτιση διαβίου σε όλη τη διάρκεια τη ζωή άσχετα με την ηλικία και τις δεξιότητες. Νομίζω ότι η έκθεση θα πρέπει επίσης να τονίζει την πρόσβαση των νέων στην αγορά εργασίας. Είναι σημαντικό. Δεν χρειάζεται να θυμίσω εδώ αριθμούς οι οποίοι πραγματικά είναι προφα... Ε, ουσιαστικά προκαλούν όλη μας την προσοχή. Απαιτείται η μεταστροφή των εργαζομένων. Οι νέοι πρέπει να μπορούν να προσληφθούν. Επίσης υπάρχει κάτι που θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε εδαφικές ανισότητες ή διαφορές. Δηλαδή, ανάλογα με τις διάφορες επαρχίες περιοχές, θα υπάρχει περισσότερη βιομηχανία, όπως ε, στη δική μου την περιοχή, στο βορρά της Γαλλίας, από ό,τι στο νότο της Γαλλίας. Αυτές οι διαφορές οι εδαφικέ, είναι κάτι που πρέπει να το θυμίσουμε και να θυμίσουμε επίση τον ρόλο των επιχειρήσεων που πρέπει να είναι και επικερδεί αλλά και να έχουν κοινωνικό πρόσωπο. Δηλαδή να επιτρέπουν ε, να δημιουργούν θέσεων εργασία χωρί να μετατοπίζονται σε άλλα φτηνότερα σημεία του πλανήτη και να δίνουν σταθερέ θέσει εργασία. Και εδώ να σταθώ σε ένα τομέα που δεν τον αναφέρουμε καθόλου, γιατί μιλάμε για ενεργειακή αποδοτικότητα. Όμω, εγώ θέλω να επιστήσω, την προσοχή σα στο εξή. Τον τομέα των κατασκευαστικών. στι οικοδομέ. Σήμερα οι οικοδομέ εκπροσωπούν το 40% των αερίων του θερμοκηπίου, το 8% του ΑΕΠ. Όλες οι μεγάλες κατασκευαστικές αύριο θα χρειαστεί να ε, αλλάξει η δραστηριότητά τους. Διότι βλέπουμε με τα κτίρια μας και βάσει τι οδηγίες που πρόσφατα εγκρίθηκε ιδίως της οδηγίας για τα κτίρια συγκεκριμένα, που λέει ότι από το 2020 μηδέν κατανάλωση ενέργειας. Λοιπόν, όλα αυτά τα κτίρια θα πρέπει να ξαναφτιαχτούν, να έχουν ενεργειακή κατανάλωση μηδέν. Άρα, η μηδενική κατανάλωση, η επισφαλής ε, ενέργεια είναι κάτι που θα επηρεάσει όλους τους επαγγελματικούς κλάδους, ε, όσους εργάζονται, τους χτίστες, τους οικοδόμους, τους, ε, ε, όλους όσους έχουν σχέση με την, κατασκευαστή, με την κατασκευή κτηρίων, όσους ασχολούνται με την αιωλική ενέργεια. Ο τομέας αυτός λοιπόν και νέες θέσεις εργασίας θα δώσει, αλλά θα πρέπει να είναι βιώσιμος και στον χρόνο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Να πάω πάλι στον εισηγητή, τον κύριο Λουμπίντσον. και μετά θα σα δώσω τι ημερομηνίε. Κύριε Λουπδίνσεν. Θα ήθελα να ευχαριστώ το, τους συναδέλφους. Λαμβάνω απόψε τις παρατηρήσεις τους στο μέγιστο βαθμό, ώστε να είναι, ώστε είναι καλή η πρόταση. Βέβαια δεν έχουμε, όπως είπα, και τόσο πολύ χώρο. Θα κάνω ό,τι μπορώ ώστε να συμφωνήσουμε στα καλύτερα αποτελέσματα. Ξέρουμε ότι δεν έχουμε να κάνουμε με ένα χώρο βιομηχανικό που ναι μεν έχει αλλάξει στον χρόνο που έχει αναμορφωθεί και που θα εξελιχθεί στο μέλλον και διαφορετικά, αλλά που εκπροσωπεί πάρα πολλέ θέσει εργασία. Ελπίζω λοιπόν ότι θα έχουμε μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Θα ήθελα απλώ να ανακοινώσω για λόγου χρονικού, Θα ξέρετε ότι έχουμε υιοθετήσει την οψευμένη διαδικασία με μία μονογλώσσα για το κείμενο. Η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 15 Νοεμβρίου Πρέπει όλες οι τροπολογίες να είναι στα αγγλικά. Ξέρω ότι αυτό θα σας δυσκολέψει, αλλά είναι ο μόνος τρόπος που είχαμε να, για να προλάβουμε τα χρονικά όρια. 15 Νοεμβρίου οι τροπολογίες, έγκριση στις 2 Δεκεμβρίου στην Επιτροπή και έτσι ολοκληρώνουμε την συνεδρίασή μας. Το απόγευμα έχουμε το ρόλο και τον αντίκτυπο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στις 3 το πρωί με, τον, με την κυρία Γκρινή.